Παρακαλώ να καθίσετε ε, όσοι στέκεστε όρθιοι πίσω. Υπάρχει χώρος επαρκής. Παρακαλώ καθίστε. Λοιπόν, θα συνεχίσω γερμανικά. Κυρίσω την έναρξη της συνεδριάσεώς μας. Το πρώτο θέμα είναι η αποδοχή της ημερησίας διατάξεως. Υποθέτω ότι δεν έχετε αντίρρηση. Και το δεύτερο θέμα είναι οι ανακοινώσει μου. Ε, υπάρχουν πολλές γλώσσες που δεν υπάρχουν σήμερα διότι δεν τις μιλάει κανείς από τους συναδέλφους όσοι θέλουν να μιλήσουν Ολλανδικά μπορούν να μιλήσουν αλλά δεν υπάρχει μετάφραση προς τα Ολλανδικά Τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης είναι η ακρόασή μας. Είμαστε πολύ ευτυχείς που μπορέσαμε να οργανώσουμε αυτή την ε, ακρόαση σήμερα κατόπιν της ετήσεως των συναδέλφων έχουμε καλέσει τέσσερις ε, ομιλητές και ομιλήτριες ένας εκπρόσωπος, ο Φέντεραλ Βάγνερ από την ε, Γερμανία, με συγχωρείτε από την Αυστρία, μετά έχουμε τον Γενικό Γραμματέα της European Cultural Foundation στο Άμστερνταμ, ο, ο οποίος ε, τώρα εγκατέλειψε τη θέση αυτή και κάνει κάτι διαφορετικό. Μετά την Κάτριν ε, Φον Βέρινγκ, η οποία ε, είναι πρώην επικεφαλής του Ευρωπαϊκού ε, Πολιτιστικού Ιδρύματος μετά τον κύριο Πολ Ντουζαντά σας βλέπω, σας βλέπω και ε, έναν συνάδελφο που τον συνοδεύει και τους ευχαριστώ που ήρθαν μετά έχουμε τον εκπρόσωπο του Φιλανδικού Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, δόκτωρ Τελίγια Ντιλικάινεν και μετά την ε, κυρία Μαρία Κοκόνεν που έρχεται από την, ε, το τμήμα της ε, κυρίας Άσφορτ στο Ευρωπαϊκό εξωτερικό, εξωτερική υπηρεσία δράσεως και έναν εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ε, καλωσορίζω όλους αυτούς. Γιατί γίνεται αυτή η ακρόαση. Ορισμένοι από εσά γνωρίζουν ότι πριν δύο χρόνια είχα οργανώσει μία ακρόαση την οποία σήμερα δεν παρίσταται αλλά δεν, δεν έγινε αυτό επίτηδες. Η είναι, είναι πολύ σημαντική. Δεν τους παρέλειψα απλώς εφόσον εργάζεται ήδη εκεί δεν υπάρχει λόγος να την ε, ξανακαλέσουμε και έτσι θέλαμε τώρα να έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με άλλους με τους οποίους δεν έχουμε ήδη συναλλαχθεί. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, γιατί ε, μας ανησυχούν οι εξωτερικές σχέσεις στον τομέα του πολιτισμού που διαδραματίζει σοβαρό ρόλο και πρέπει γιατί αυτό σημαίνει πώς συνειδητοποιούμε τον κόσμο και συμβάλλει στον διαπολιτιστικό διάλογο βέβαια. Προσπαθούμε όπου έχουμε πολιτιστικές σχέσεις να εξασφαλίσουμε ε, την πρόοδο και την εξέλιξη, πράγμα το οποίο επιτυχάνεται διότι έτσι ενισχύουμε τα ανθρώπινα ονόματα και έχουμε και άλλες ε, δυνατότητες όπως το έχουμε δει ε, στα Δυτικά Βαλκάνια παραδείγματο χάρη και το χρειαζόμαστε. Δηλαδή ο πολιτισμός στηρίζει την κοινωνία των πολιτών και ίσως ε, κάτι άλλο το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερος συναδέλφους είναι θέμα οικονομικής εξελίξεως. Δεν θέλουμε να παραβλέψουμε ούτε αυτή την παράμετρο. Οπότε θα έπρεπε ήδη για τα υπάρχοντα δίκτυα τα οποία δραστηριοποιούνται όπως η ΟΗΝΙΚ παραδείγματος χάρη να τα στηρίζουμε διότι πρόκειται για πολιτιστικά Ινστιτούτα τα οποία έχουν ε, δραστηριοποιηθεί στην ΟΗΝΙΚ όπως το Ινστιτούτο Γκέτε, μετά μέσω της UNESCO με την Επιτροπή του, από το 2005 τα κράτη-μέλη της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως έχουν δεσμευτεί να θεωρήσουν τον πολιτισμό σαν βασικό τομέα των εξωτερικών τους σχέσεων ε, και να προωθήσουν τις διεθνείς σχέσεις στον τομέα αυτό. Είναι ε, θαυμάσια λόγια, ε, έχουν προσυπογραφεί, αλλά το εάν ακόμη εφαρμόζονται είναι κάτι που πρέπει να επαληθεύσουμε και έχει γίνει και ε, ένα ψήφισμα από την συνάδελφο Σάκε ε, για τα θέματα αυτά και σε αυτό ε, το ψήφισμα λέγεται ότι όλα τα θεσμικά όργανα πρέπει να θεωρήσουν ότι ο πολιτισμός είναι ε, βασική πτυχή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και έτσι ε, και αυτό, ε, αυτή η ακρόαση είναι ένα λιθαράκι προς αυτήν την κατεύθυνση. Όπως σας το περιέγραψα θα προχωρήσουμε τώρα. Έχουμε τέσσερις τέσσερις ε, ηθήνοντες οι οποίοι θα μπορέσουν να λάβουν το λόγο επί πέντε λεπτά και μετά θα ελπίζω ότι θα υπάρξει ένας διάλογος και μετά οι εμπειρογνώμονες αυτοί θα έχουν πάλι πέντε λεπτά έκαστος για να εκφραστούν και μετά θα δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο. Ε, θέλω να σας πω και να σας επισημάνω και ένα τεχνικό θέμα διότι υπάρχει μετάδοση στο διαδίκτυο αυτής της συνεδριάσεων. Βέβαια βλέπουμε τα άδεια έδρανα αλλά δυστυχώς δεν μπορώ κάτι να κάνω. Το έχω πει στους συναδέλφους ότι υπάρχει web streaming, δηλαδή μπορεί ο, κάθε ψηφοφόρος να παρακολουθήσει τι γίνεται στο Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρακαλώ λοιπόν να ε, ε, να ε, χρησιμοποιείτε πάντοτε το μικρόφωνο που είναι αριστερά σας για να μπορέσει να στραφεί η κάμερα και μετά να σβήσετε το κουμπάκι για να μπορέσει να λάβει το λόγο επόμενος. Δίνω λοιπόν τον πρώτο, στον πρώτο το λόγο στον κύριο Βάγνερ σε οποιαδήποτε γλώσσα επιθυμεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ντόρις Πάκα, κυρία Πρόεδρε, Πρόεδρε της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής αυτής και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την ε, εισηγήτρια της σημαντικής αυτής έκθεσης, την κυρία Σάκη. θα μιλήσω εκπροσωπώντα την κοινωνία των πολιτών, ότι εργάζομαι αυτή τη στιγμή στη Βιέννη στο Υπουργείο Πολιτισμού. Πάντω η κοινωνία των πολιτών με βοηθάει πολύ στην ιδιαίτερη αυτή αποστολή, στη ιδιαίτερα καθήκοντα τα οποία έχω. Και θα ήθελα σήμερα να παρουσιάσω μία πρωτοβουλία των πολιτών που ονομάζεται More Europe, Περισσότερη Ευρώπη, και που έχει ω στόχο να εμπλουτίσει περισσότερο με πολιτισμικά θέματα την πολιτική εξωτερικών σχέσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα μιλήσουμε σήμερα για την υλοποίηση, την εφαρμογή προτάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να ξεκινήσω όμως με δύο βασικές έννοιες. Καταρχάς, αναφερόμαστε όλο και περισσότερο στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, ακόμα και στον τομέα αυτό του πολιτισμού, που έχει να κάνει με δημιουργικές βιομηχανίες, που έχει να κάνει με σχετικές αγορές, που έχει να κάνει με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ασχολούμαστε και με το ζήτημα της συνεργασίας, γιατί η σύγχρονη πολιτιστική διπλωματία έχει να κάνει με το να ακούμε και να συνεργαζόμαστε καλύτερα με τους εταίρους μας. Δεύτερη παρατήρηση. Τη στιγμή αυτή που δημιουργεί σιγά σιγά η Ευρωπαϊκή Ένωση μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ακόμα μια συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά την πολιτισμική πολιτική. Και αν δούμε τις μεγάλες δυνάμεις του παρελθόντος, του παρόντος, αλλά και τις αναδυόμενες ε, δυνάμεις του μέλλοντος, θα δούμε πόσο μεγάλη σημασία δίνουν στη λεγόμενη soft power, στην ήπια αυτή δύναμη, στην πολιτισμική διπλωματία. Ας δούμε για παράδειγμα την χρήση που έχουν κάνει οι Ηνωμένε Πολιτείε στο παρελθόν, αλλά και τη χρήση που κάνει τώρα η Κίνα που είναι μια πολύ σημαντική αναδυόμενη οικονομία και η οποία έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί πάρα πολύ τα νέα τεχνολογικά μέσα, όπως για παράδειγμα τους υπολογιστές και πώς έχει εμπλουτίσει ουσιαστικά την εξωτερική της πολιτική με την πολιτισμική αυτή πολιτική, με διάφορα πολιτισμικά μέσα. Ας επανέλθω τώρα στην πρωτοβουλία μας More Europe, περισσότερη Ευρώπη. Είμαστε μια πρωτοβουλία των πολιτών, της κοινωνίας των πολιτών γιατί ουσιαστικά πολιτισμός αποτελεί ένα πολιτισμικό σχέδιο. Η ονομασία «Περισσότερη Ευρώπη» φαίνεται ιδιαίτερα παράδοξη, τη στιγμή που φαίνεται ότι καταραίει σιγά-σιγά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε για αυτό το λόγο να εμφυσίσουμε νέα εμπιστοσύνη στα πλαίσια της κοινωνίας των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και προς α, τις τρίτες χώρες. Θέλουμε ουσιαστικά να λειτουργούμε διαφορετικά στο παγκόσμιο προσκήνιο, στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης. Πρόκειται λοιπόν για μια πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να αντιταχθεί σε αυτό, τον, αυτό το κοινικό κίνημα καταστροφής το οποίο βλέπουμε τελευταία. Θέλουμε να συνεργαζόμαστε περισσότερο, να επενδύσουμε περισσότερο στον διαπολιτισμικό διάλογο παγκοσμίω. Κυρίε και κύριοι, προφανώ εσεί γνωρίζετε πολύ καλά τα πάντα σχετικά με το soft power, με την ήπια δύναμη, την ήπια εξουσία. Έχετε παράγει μια πολύ σημαντική έκθεση που αποτελεί βάση για μα και είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι θα πρέπει να κάνουμε τόσο στο παρόν όσο και στο άμεσο μέλλον. Στα πλαίσια της διαδικασία λοιπόν αυτής πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες. Αυτό έχει να κάνει τόσο με την εργασία που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την αντίστοιχη Γενική Διεύθυνση, όσο και με την εργασία που κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και με την εργασία που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική και Δράση. Δεν ακούγεται όμω αρκετά η φωνή των πολιτών. Οι πολίτε θέλουν μια πιο ισχυρή Ευρώπη. Υπάρχουν δημοσκοπήσει που το καταδεικνύουν αυτό. Πιστεύουμε όμω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί περισσότερο αυτή η διαπολιτισμική συνεργασία. Αυτό το soft power θα πρέπει να εμπεριέχεται περισσότερο στις μελλοντικέ πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να εμπλακούν περισσότερο οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, η κοινωνία των πολιτών στην πολιτική που θα ακολουθηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια εντελώς νέα πολιτική. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ακούσετε τους πολίτες και έχουμε κάποια πολύ θετικά παραδείγματα, κάποια αποδεικτικά στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν ότι πρέπει να επενδύσει περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον στην πολιτισμική διπλωματία, την δημόσια διπλωματία και θέλουμε ουσιαστικά την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει εμεί στον τομέα αυτών να τη μοιραστούμε μαζί σα. Είμαστε ακόμα μια μικρή ομάδα που ασκεί όμω σημαντική επιρροή. Στη βάση μας έχουμε το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Ίδρυμα, καθώς επίσης και άλλα ιδρύματα, άλλα Ινστιτούτα, καθώς επίσης και ε, ε, πολύ σημαντικούς εταίρους από την κοινωνία των πολιτών. Θέλουμε λοιπόν να συνεργαστούμε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσα στο επόμενο αυτό χρόνο. Πρόκειται για ένα νέο σχέδιο, δεν πρόκειται για μια νέα δομή, γιατί τη δομή την έχουμε ήδη, είναι το UNIC. Είναι τα εθνικά, πολιτιστικά Ινστιτούτα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα θέλαμε λοιπόν να πετύχουμε συγκεκριμένους στόχους μέσα στο επόμενο έτος ένας μικρός ε, αριθμός πολιτιστικών Ινστιτούτων με σημαντική εμπειρία έχουν αποφασίσει να μας ε, βοηθήσουν το Βρετανικό Συμβούλιο, το Γαλλικό Ινστιτούτο, το Institut Français, το Γερμανικό Ινστιτούτο ΙΦΑ, καθώς επίσης και το Δανέζικο Ινστιτούτο, καθότι η, Δανέζικη, η Δανία θα έχει την Προεδρία του χρόνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα θέλανε λοιπόν αυτά τα πολιτιστικά Ινστιτούτα να κάνουν το ακόλουθο. πρώτο, να δημιουργήσουν ε, έναν έντονο διάλογο, έντονε συζητήσει και επίσης να καταφέρουν να προσωπήσουν καλύτερα την πολιτική μας αυτή. Χρειαζόμαστε τα απαραίτητα πλέον μέσα. Δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε απλώς μόνο για εξωτερικές σχέσεις και πολιτισμό, πρέπει να αρχίσουμε να ελοποιούμε τα λόγια μας αυτά. Χρειάζονται λοιπόν οι απαραίτητες δομές, η απαραίτητη συντονιστική δομή που θα καταφέρει να συντονίσει τις προσπάθειες που γίνονται από τα διάφορα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα διάφορα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Θέλουμε επίσης να συντονίσουμε καλύτερα την εθελούσια προσπάθεια των πολιτιστικών Ινστιτούτων των κρατών μελών. Θέλουμε να καταφέρουμε να προσελκύσουμε τους απαραίτητους πόρους και τέλος θέλουμε να δημιουργήσουμε την απαραίτητη στρατηγική που θα βασίζεται στην, στο να αφουγκραστούμε ουσιαστικά καλά τις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ορατή στρατηγική αυτή τη στιγμή και ελπίζουμε ότι σε ένα χρόνο θα έχουμε καταφέρει να έχουμε μία δομή συντονισμού που θα καθιστά ουσιαστικά τα κράτη-μέλη πολύ καλύτερους συνομιλητές της κοινωνίας των πολιτών και των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών. Και θα καταφέρουμε, πιστεύω, να πετύχουμε το αποτέλεσμα αυτό τόσο στα μεγάλα όσο και στα μικρά κράτη-μέλη. Είναι πολύ σημαντικό να ακούμε και τις μικρές χώρες κάθε φορά που θεσπίζουμε στόχους πολιτικής. Θα πρέπει λοιπόν να συνομιλήσουμε με αυτού οι οποίοι έχουν πολύ σημαντική επιρροή, να μιλήσουμε και με αυτού που εργάζονται στα μέσα ενημέρωση. Έτσι λοιπόν στι πρωτεύουσε τη Ευρώπη τα επόμενα χρόνια θέλουμε ακριβώ να δημιουργήσουμε αυτή την έντονη συνεργασία προκειμένου να καταφέρουμε να ευαισθητοποιήσουμε του ηθήνοντε για ζητήματα πολιτική, αυτού που χαράσουν πολιτική εντό και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά όσον αφορά την ε, συζήτηση που πρέπει να γίνει. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι μορφή θα πρέπει να πάρει στο μέλλον. Έχουμε κάποια επιτυχημένα εργασία, εργαλεία με σε επίπεδο κρατών μελών. Έχουμε τα απαραίτητα δίκτυα πολλές φορές μέσω καλλιτεχνικών σχολών κτλ. Δεν ξέρουμε όμως ποια μορφή θα πάρει κοινή προσπάθεια στο τέλος. Θα έχουμε ένα Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τους ε, Ευρωπαϊκούς ε, Πολιτισμούς, θα καταφέρουμε να έχουμε μια γενικότερη υποστήριξη, θα έχουμε ε, εντεταλμένους για πολιτιστικά θέματα σε διάφορες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή προσπαθεί να δει τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να γίνει και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, αν υπάρχουν κάποια περιθώρια για τη λεγόμενη πολιτισμική διπλωματία. Πάντως, σε κάθε περίπτωση η τελική δομή θα πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό το λόγο πηγαίνουμε σε πόλεις όπως το Λονδίνο, το Παρίσι, το Βερολίνο, το Άμστερνταμ, η Κοπενχάγη και προσπαθούμε εκεί σε τοπικό επίπεδο να συζητήσουμε με τους ηθήνοντες, με τα μίντια, με τα ενδιαφερόμενα μέρη και επιστρέφουμε έπειτα στις Βρυξέλλες για να αποφασίσουμε. Στα πλαίσια λοιπόν της πρωτοβουλία μας διοργανώσαμε μια συζήτηση με τους επικεφαλής ε, της, θα όργανώσουμε μάλλον μια συζήτηση με τους επικεφαλείς της Unix της Βρυξέλλης στις 8 Δεκεμβρίου και ελπίζω ότι θα καταφέρω να σας αποκαλύψω τότε περισσότερα μυστικά από αυτά τα οποία σας λέω τώρα. Θα θέλαμε πάντως να συνεργαστούμε και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την κυρία Χά και την εισηγήτριά σας καθώς επίσης και με την επικεφαλής της Επιτροπής Πολιτισμού και ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να σας βοηθήσουμε να βγείτε κι εσείς λίγο από τις Βρυξέλλες, να απομακρυνθείτε από τις Βρυξέλλες και να δραστηριοποιηθείτε περισσότερο σε τοπικό επίπεδο στη συζήτηση αυτή που διοργανώνουμε. Συζητήσεις λοιπόν, έντονες συνεργασίες με τους ηθήνοντες, θέλουμε να καταλήξουμε στην απαραίτητη δομή, στους απαραίτητους πόρου που θα μας επιτρέψουν να έχουμε τον απαραίτητο συντονισμό, την απαραίτητη αλληλοσυμπληρωματικότητα, να απομακρυνθούμε περισσότερο από τη γραφοκρατία και να έχουμε μια ξεκάθαρη στρατηγική, μια ορατή στρατηγική. Νομίζω ότι ανάλωσα άλλο το χρόνο που με αναλογούσε. σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Νομίζω ότι χαίρεται πολύ ότι υπάρχει αυτή η εξωτερική βοήθεια η οποία μπορεί να οδηγήσει στα σωστά συμπεράσματα. Δεν το άκουσε αλλά θα το επαναλάβουμε. Και τώρα η Κατερίνα Ντίτριχ. για να έχουμε ένα πιο έντονο πολιτιστικό στοιχείο στην ευρωπαϊκή πολιτική. Θα πρέπει να αποδείξουμε στον εξωτερικό κόσμο πως η, η μία εξωτερική πολιτιστική πολιτική και η πολιτιστική ευρωπαϊκή πολιτική αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Στο εσωτερικό έχει να κάνει με την προστασία της ποικιλομορφίας των πολιτισμών μας, που αποτελεί ένα από τα ε, αναπόσπαστα συστατικά της διαδικασίας ολοκλήρωσης της Ευρώπης και σε εξωτερικό επίπεδο έχει να κάνει με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα πολιτιστικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που θα ενώσουν την Ευρώπη και θα, και θα δημιουργήσουν ένα ευρωπαϊκό έργο το οποίο θα σέβεται κοινέ πεπιθήσεις και αξίες. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να θεωρηθούμε απειλή για τον κόσμο εκτός Ευρώπης. Θα πρέπει λοιπόν να συντονίσουμε και να ευθυγραμμίσουμε αυτή τη στιγμή τις κατακαιρματισμένες εξωτερικές πολιτικές και τα project της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί συμπεριλαμβάνουν ε, ένα συστατικό ε, στοιχείο πολιτιστικό και επίσης θα πρέπει να προωθήσουμε τα πολιτιστικά έργα σε τρίτες χώρες ε, σε συνεργασία με τα υφιστάμενα δημόσια και ιδιωτικά πολιτιστικά δίκτυα. Προτείνω λοιπόν τα εξής εργαλεία, δράσεις και μέσα. Δεν είναι κάτι το επαναστατικό ή προκλητικό γιατί τα περισσότερα ήδη υπάρχουν αλλά δεν μοιάζουν να είναι υπαρκώς συντονισμένα και δεν θεωρώ πως, όπως μπορούν να κρυθούν υπαρκώς ορατά. Θα πρέπει λοιπόν να εντάξουμε ένα συντονιστικό ε, τμήμα στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης που θα αναλάβει τις εξής αρμοδιότητες και αναφέρομαι σε κάποιες από αυτές. Θα συνεδριάζει σε τακτικά χρονικά διαστήματα με εκπροσώπους άλλων γενικών διευθύνσεων ε, των οποίων οι πολιτικές συμπεριλαμβάνουν μια πολιτιστική διάσταση. Εξωτερική, εμπορική, διεύρυνση, δράση για το κλίμα, ανάπτυξη, πολιτισμό και παιδεία για παράδειγμα. Και θα υποβάλουν μία ή δύο φορές το χρόνο μία έκθεση για τα αποτελέσματα αυτής της δράσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, θα πρέπει τα αποτελέσματα αυτών των συναντήσεων να γίνουν πιο ορατά για τους ε, ετούντες και για όσους ε, επιχορηγούνται σε μία ιστοσελίδα, σε έναν ιστότοπο ε, στα αγγλικά, όπου θα ενημερώνεται συνέχεια. Γιατί βέβαια υπάρχει μία, ένας γερμανικός ιστότοπος που λέγεται Europa for Third Culture ε, και αναφέρεται και συγκεκριμένα στη συνεργασία με τρίτες χώρες, έχει βέλτιστες πρακτικές κτλ. Δεν είναι κάτι λοιπόν το καινούριο. Η αρχική εκδοχή ήταν γαλλική ε, και έχουμε και μία γερμανική, οπότε χρειαζόμαστε και κάτι στα αγγλικά, μία διευρυμένη εκδοχή που θα αναφέρεται στα ορατά αποτελέσματα. Μπορούμε επίσης να επεκτείνουμε και έναν ιστότοπο ο οποίος ήδη υφίσταται, που είναι το Εργαστήριο για την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Συνεργασία, που καλύπτει όλα τα ευρωπαϊκά ε, πολιτιστικά έργα συνεργασίας σε τρίτες χώρες. Θα μπορούσε και αυτό να γίνει. Όλα αυτά είναι υπηρεσίες ενημέρωσης και πληροφόρησης, οι οποίες απλώς θα είναι πιο συντονισμένες. Θα πρέπει όμως να δημιουργηθεί και ένα πλαίσιο αναφοράς που θα στηρίζει τα άξια στήριξης έργα ε, πολιτιστικής συνεργασίας σε τρίτες χώρες με μία αυξανόμενη συλλογή βέλτιστων πρακτικών, γιατί υπάρχουν αρκετές και έχουν περιγραφεί. Υπάρχουν παντού αλλά δεν έχουν συλλεχθεί σε μια βάση. Δεν έχουν συγκεντρωθεί και είναι δύσκολο να δημιουργηθεί στη θεωρία αυτό το πλαίσιο αναφορά, γιατί η κατάσταση είναι διαφορετική στα διάφορα κράτη. Αλλά αν έχουμε 100-150 παραδείγματα, τότε νομίζω πω η κατάσταση θα είναι πιο ξεκάθαρη. Θα πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε ε, δημιουργώντας ένα μικρό ταμείο προσαρμογής για την συμπερίληψη ε, των μικρότερων και ασθενέστερων οικονομικά μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στα σχέδια συνεργασίας σε Πολιτική συνεργασία με, τρία, με τρίτα κράτη και να δημιουργήσουμε και ένα συνδεδεμένο πανευρωπαϊκό πρόγραμμα επισκεπτών για τα μεγάλα κράτη, το οποίο θα αποδείξει πως σεβόμαστε την αρχή της αλληλεγγύης, κάτι το οποίο θα χρησιμοποιηθεί και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξωτερικά. Μπορούμε λοιπόν να στηρίξουμε την πρωτοβουλία Περισσότερη Ευρώπη, More Europe, και να διατηρήσουμε μια τακτική ανταλλαγή ιδεών με την Προεδρία της ε, Ιουνής, όπως επίσης και με το γραφείο του στο συντονιστικό στις Βρυξέλλες, έτσι ώστε να προωθήσουμε μελλοντικά ε, έργα πολιτικής συνεργασίας σε τρίτες χώρες και να μπορέσουμε να ε, συλλέξουμε βέλτιστες πρακτικές. Και αν κοιτάξετε τον ιστότοπο της Ιούνης θα δείτε πως όντως εκεί έχουν συμπεριλάβει κάποια τέτοια παραδείγματα. Εκπαίδευση θα πρέπει σε κάθε ε, αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρίτες χώρες ένας αξιωματούχος να είναι υπεύθυνο για τα πολιτιστικά και να εκπαιδευτεί για το έργο αυτό. Και αυτό θα μπορούσε να γίνει, ε, να είναι η αποκλειστική αρμοδιότητα ή να θεωρηθεί μια αρμοδιότητα ανάμεσα σε άλλες για τον ή την αξιωματούχο αυτή ή αυτόν ε, και ίσως δίνοντας και κάποια προώθηση στη συνεργασία με άλλα προγράμματα κατάρτισης, για παράδειγμα αυτό της Γιούνης. Επίσης, θα πρέπει να κάνουμε λόμπινγκ στις επιτροπές νομικών θεμάτων, οικονομικών θεμάτων για τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι τέχνες και ο πολιτισμός τη στιγμή της προετοιμασίας νόμων και της κατανομής κονδυλίων. Δηλαδή να υπάρχει μια ρήτρα, για παράδειγμα, προσαρμοστικότητας, λήψης υπόψη των πολιτιστικών διαστάσεων κτλ. Κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν σας αποκαλύπτω και νομίζω ότι θα με πιστέψετε γιατί υπάρχουν τρεις σχετικές μεγάλες μελέτες που αποδεικνύουν ε, μαζί με αυτήν ε, που σηκώνω, γιατί έχω μόνο ένα αντίγραφο, δεν μπορώ να σας το δώσω ένα αντίτυπο, αλλά είναι στα αγγλικά και στα γερμανικά, που αποδεικνύουν πως πως οι δημόσιοι παίκτε σε όλα τα κράτη-μέλη, σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι μεγάλοι πολιτιστικοί παίκτε, από του οποίου ζητήθηκε η γνώμη. Όπως επίσης, ούτε τα ιδιωτικά δίκτυα θα έφεραν αντίρρηση για οποιαδήποτε τέτοια συντονισμένη εξωτερική πολιτική, η οποία θα συμπλήρωνε, και το λέω αυτό, δεν μπορώ να το τονίσω αρκετά, που θα συμπλήρωνε και θα ενίσχυε όλη αυτή τη συνεργασία που γίνεται σε ε, τοπικό και περιφερειακό ε, επίπεδο για θέματα πολιτισμού στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρον και ε, πολλά στοιχεία που δεν είναι καινούρια αλλά ορισμένα δεν έχουν προχωρήσει. Και τώρα θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Τζουζαντά από τον Μποζά στις Βρυξέλλες να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ ε, κυρία Πρόεδρε και μέλη της Επιτροπής που, για την πρόσκληση αυτή. Ο συνάδελφός μου Φρεντερίκ Μιουζέ που είναι συν υπεύθυνο ε, στο Μποζάρ έχει δημιουργήσει μέσα στο ε, κτίριο του Μποζάρ ε, μία υπηρεσία και θα δείτε εδώ την ιστορία του κτηρίου αυτό το οποίο ήταν κάτω από τον χώρο της καγκελαρίας στο Βέλγιο και από τις ε, ε, δημιουργίες του μετά το τέλος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου ε, συνέβαλε στη δημιουργία της κοινωνίας των πολιτών στη δεκαετία του 20 μετά το, όπως είπαμε το τέλος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Έχουμε μία διμερή συνεργασία με το πρόγραμμα Ευρωπαλία το οποίο προσπαθήσαμε να κάνουμε πιο πολυμερές και ε, δημιουργήσαμε το Passage to Asia επί τη ευκαιρία της συνεδριάσεως των ΑΣΕΜ ε, και επιτρέψαμε ενισχυμένες επαφές μεταξύ του Βελγίου, των ευρωπαϊκών χωρών ε, και περισσότερη πολιτιστική ε, διπλωματία. Υπάρχουν, ε, ε, υπάρχουν μεν πρωτοβουλίες αλλά στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας πρέπει να τις αναπτύξουμε διότι υπάρχει μία ανάπτυξη της cultural diversity και επίσης η συμμετοχή για τις ε, ε, για ε, διάφορες εκδηλώσεις όπως η Media Mundi με τις χώρες ΣΑΚΕ και το 2009 δημιουργήσαμε μία νέα στρατηγική η οποία όμως δεν έχει εξελιχθεί ακόμη. Ε, από το 2007 έχουμε 200 εκατομμύρια ευρώ που έχουν αποδοθεί για πολιτιστικά προγράμματα στις ε, τρίτες χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ε, δεν επαρκούν και όλα αυτά εξαρτώνται και από συζητήσεις πολιτικές σε υψηλό επίπεδο και δεν μπορεί κανείς έτσι να προωθήσει και να περιλάβει τον πολιτισμό σε ένα διεθνές πρόγραμμα διότι είμαστε σε έναν κόσμο πολύ πολιτιστικό και υπάρχουν μετακινήσεις και συναντήσεις μεταξύ των λαών υπάρχει δηλαδή μεγαλύτερος ρόλος των κέντρων τέχνης σαν το Μποζουάρ για να ενισχύσουν το διάλογο μεταξύ των κοινωνιών και των υπήρων και να προωθήσουν τη δημιουργικότητα. Είναι ένας θαυμάσιος ρόλος ε, με το know-how προς τις τρίτες χώρες ε, διότι η τέχνη είναι βασικός ε, τρόπος για να κατανοήσουμε τους άλλους και αποτελεί ένα βασικό στοιχείο της διπλωματίας στο σημερινό κόσμο και άρα πρέπει να προωθήσουμε την ε, πολιτιστική διπλωματία διότι μόνο έτσι μπορούμε να προωθήσουμε τις αξίες μας και για να μπορέσουμε να προωθήσουμε βασικές αξίες και ε, σας παραθέτω την φράση του Χαβιέ Σολάνας που είναι πολύ σχετική με το θέμα μας. Δηλαδή η Ευρώπη δεν μπορεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνη της. Μπορούμε να ανοίξουμε μεν πρωτές προς ε, τις ε, τρίτες χώρες βάσει βάση της εμπειρίας που έχουμε και παραδείγματο χάρη με το πρόγραμμα όραμα για την Αφρική με εκθέσεις, με θέατρα και το Μποζάρ λειτουργεί ε, σαν πρέσβη σήμερα για να ενισχύσουμε μία σαφή εικόνα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ανά τον κόσμο, μία εικόνα που ήδη υπάρχει και ο πολιτισμός και οι συμμετέχοντες σε αυτόν παρουσιάζονται διεθνώς και αυτό είναι πολύ πιο προφανές εκτός Ευρώπης από ό,τι εντός διότι ο κόσμος αξιολογεί την Ευρώπη βάσει των πολιτιστικών της αξιών. Συνεργαζόμαστε με την Αίγυπτο στα πλαίσια του, του Μποζάρ για την περίοδο 2012-2014 για να μπορέσουμε να προσθέσουμε τα στοιχεία του 21ου αιώνα αλλά και ε, την ε, ε, πορεία της ιστορίας του παρελθόντος για την κοινωνία των πολιτών, για την επικοινωνία, για να παρουσιάσουμε μία διαφορετική εικόνα της Αιγύπτου. Έχουμε ξεκινήσει πριν από την Επανάσταση και θέλουμε να δείξουμε κάτι παραπάνω από τις πυραμίδες και τις καμήλες που είχαμε στο παρελθόν να μπορέσουμε σήμερα να δείξουμε πως ε, η τέχνη στήριξε την κοινωνία και αποτέλεσε μία ήπια δύναμη για να μπορέσει να προωθήσει τη συνεργασία σε όλη την Μεσόγειο και είναι μια δυνατότητα για να παρουσιάσουμε τον ρόλο του στοιχείου αυτού σε μια περίοδο κρίσεως μακριά από τους πολιτικούς και ε, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και μία σύσταση την οποία έχουμε κάνει, δηλαδή ε, πώς ε, θα μπορέσουμε να καταρτήσουμε αυτή την εξωτερική πολιτιστική πολιτική τη συνεργασία με τρίτες χώρες που πρέπει να ενταχθεί σε ένα σύνολο με τη ε, συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της κυρίας Άστον και να υπάρχει μία εγκάρσια επίδραση σε όλες τις εξωτερικές πολιτικές οριζοντίως και περιφερειακά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Καλύτερη συνεργασία με τρίτες χώρες μέσω των πρεσβειών, των δικτύων της κοινωνίας των πολιτών και των πολιτιστικών κέντρων για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τις κινήσεις αυτές σε ε, ξένες ε, χώρες και ακούσαμε πολλά από αυτού σήμερα το απόγευμα ήδη. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ε, ε, τονίσουμε περισσότερο το στοιχείο των ε, πρέσβεων για να μπορέσουμε να προβάλλουμε όλα τα στοιχεία προς τα έξω και της πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και των ζωντανών τεχνών και της κοινωνία των πολιτών, τη θέση της γυναίκας στην Αίγυπτο, στην Τουρκία, ε, να ε, περιλάβουμε την επικοινωνία και όλες τις γλωσσικές πτυχές ε, και όλα αυτά τα θέματα να αναπτυχθούν περισσότερα. Έχω αυτές τις πέντε συστάσεις τις οποίες απευθύνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο ε, Τάγια Τιλικάινερ από το Φιλανδικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη της ε, Επιτροπής, Νομίζω ότι ε, η έκθεση της εισηγήτριάς σας είναι ιδιαίτερα πλήρης και συμφωνώ απόλυτα με τα βασικά σημεία εκκίνησης ε, πολιτικής φύσης της έκθεσης αυτής. Για παράδειγμα, πως διαβάζω ότι θα πρέπει να ενδυναμωθεί η ε, ταυτότητα της ε, Ευρώπης, η πολιτιστική ταυτότητα της Ευρώπης, ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί περισσότερο ο πολιτισμός στην επίτευξη διάφορων πολιτικών στόχων και καθότι καθότι διαμορφώνονται νέε συνθήκε γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και καθότι τρίτε χώρε χρησιμοποιούν περισσότερο την έννοια του soft power, ανάλογη δράση θα πρέπει να αναλάβει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει ο πολιτισμό να αποτελέσει αναπόσπαστο στοιχείο τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και τη εξωτερική πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να αναφερθούμε περισσότερο στον ρόλο που θα μπορέσει να διαδραματίσει η πολιτιστική διπλωματία, με συγχωρείτε, ιδίω στα πλαίσια τη δράση που θα αναλυφθεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Θα πρέπει να προωθηθεί περισσότερο το ευρωπαϊκό μοντέλο. Στο παρελθόν υπήρχε ένα μεγάλο ενδιαφέρον για το ευρωπαϊκό αυτό μοντέλο Υπήρχαν διάφορα στερεότυπα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η πολιτική που ακολουθεί ουσιαστικά επιλύει ειρηνικά τις διάφορες διενέξεις, ότι ακολουθείται μια περιεθνική διακυβέρνηση, ότι ακολουθείται ένα μεταβεσθαλικό μοντέλο όσον αφορά την υπηκότητα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπήρχε ένα πολύ μεγάλο ε, διεθνέ ενδιαφέρον για τα χαρακτηριστικά αυτά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τα χρησιμοποιεί άραγε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το ερώτημα και εγώ εκφράζω κάποιε αμφιβολίες. Θα μπορούσαμε λοιπόν να δούμε περισσότερο πώς θα καταφέρουμε να χρησιμοποιήσουμε την πολιτιστική συνιστόσα των εξωτερικών σχέσεων, προκειμένου να καταφέρουμε να προωθήσουμε περισσότερο το ευρωπαϊκό μοντέλο, το παλιό ευρωπαϊκό μοντέλο προς τα έξω. Στην έκθεση γίνεται αναφορά στον πολιτισμό ως μέσο για την ε, ηρωνική διευθέτηση των ε, διεθνών σχέσεων. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό συνάδει πολύ καλά με την προώθηση του ευρωπαϊκού μοντέλου μέσω του πολιτισμού. Ποια πολιτιστικά μέσα θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, μέσω ποιων πολιτισμικών μέσων θα μπορούσαμε ουσιαστικά να προωθήσουμε το ευρωπαϊκό μοντέλο ολοκλήρωσης. Τρεις συγκεκριμένε προτάσεις θα ήθελα να κάνω. Θα πρέπει να δούμε αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο διάφορα έργα, ταινίες, ντοκιμαντέρ, προκειμένου να καταφέρουμε να έρθουμε πιο κοντά στους πολίτες και να αναφερθούμε περισσότερο, να διαφημίσουμε περισσότερο την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Την όλη διαδικασία συναπόφασης που βρίσκεται πίσω από το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, να αναφερθούμε σε κάποιες βασικές ηγετικές φυσιογνωμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βοήθησαν πάρα πολύ την ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα έξω, προς το γενικότερο ευρύτερο κοινό θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσουμε τα διάφορα συστήματα συνεργασίας που υπάρχουν μεταξύ σχολείων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τα συστήματα ανταλλαγής καθηγητών. Θα μπορούσαμε να εμπλουτίσουμε το πρόγραμμα αυτό με την ανταλλαγή, με τον εμπλουτισμό μάλλον του διδακτικού υλικού. Στην έκθεση γίνονται κάποιες σχετικές προτάσεις και τις χαιρετίζουν. Επίσης, Είμαι υπέρ τη διεύρυνση του δικτύου ευρωπαϊκών σποδών. Έχουμε το σύστημα Ζαμονέ, το οποίο έχει να κάνει με την ακαδημαϊκή έρευνα και το οποίο μας βοήθησε ιδιαίτερα στο να διαδώσουμε περισσότερο το ευρωπαϊκό μήνυμα μέσω των πανεπιστημίων, τόσο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω λοιπόν ότι το σημαντικό αυτό υφιστάμενο σύστημα θα μπορούσε να εμπλουτιστεί περισσότερο και να χρησιμοποιηθεί και από διάφορα ε, ερευνητικά ιδρύματα και think tanks και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα βοηθήσει λοιπόν και η ιδέα αυτή να καταστήσουμε το ευρωπαϊκό παράδειγμα πιο ορατό, να το προωθήσουμε περισσότερο. Το ευρωπαϊκό μοντέλο δηλαδή για την διακυβέρνηση, για την επίλυση των διευθετήσεων, για την ε, έννοια της μεταβεσφαλικής υπηκότητας. Είναι ε, μοναδικά χαρακτηριστικά αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αξίζει να προωθήσουμε περισσότερο προς τα έξω. Δεν θα ήθελα τώρα να επαναλάβω πράγματα τα οποία είπαν οι συνάδελφοι. Θα ήθελα να επιμείνω στο ότι πιστεύω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε κάπως περισσότερο στις προτάσεις που γίνονται στην έκθεση, αλλά και να δούμε πού θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο την, την πολιτιστική διπλωματία. Αυτό είπαν άλλωστε και οι προαλήσαντες, να καταφέρουμε να εντοπίσουμε περισσότερες ευκαιρίες χρησιμοποίησης της πολιτισμικής διπλωματίας και πέρα από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Έχουμε, όπως βλέπω εδώ πέρα, τα κατάλληλα μέσα προκειμένου να διευρύνουμε περισσότερο το μήνυμα αυτό. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν περισσότερο, πιστεύω, την πολιτιστική διπλωματία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Ε, έχω μία παρατήρηση αλλά τώρα θα συγκρατηθώ και δεν θα την κάνω. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι εδώ έχουμε και την Κρίστα Μπρίτς που η οποία ήταν ε, σε αυτή την επιτροπή και η οποία έχει κάνει πολλά ε, μαζί με την ε, Helga Τρίπελ και μαζί μου και τώρα είναι νοικοκυρά στη, πίσω στην πατρίδα της. Χαίρομαι και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να σε χρησιμοποιήσουμε σαν εμπειρογνώμονα. Δυστυχώς όμως μπορούμε να έχουμε μόνο δύο ο εμπειρογνώμων ε, Χαίρομαι ε, που ε, έμεινε τώρα, ότι έμεινες εδώ για κάποιο χρονικό διάστημα και τώρα δεν κατάφερες να επανεκλεγείς την τελευταία φορά. Δεν ξέρουν δηλαδή οι περισσότεροι ψηφοφόροι στις χώρες πόσο προσπαθούμε. Αλλά τώρα έχω να δώσω το λόγο και σε κάποιον ακόμη και αυτό είναι η εκπρόσωπος της κυρίας Άστον, η κυρία Μαρία Κοκόνεν. Πού είναι? Ε, μάλιστα. Εγώ έψαχνα αλλού. Με συγχωρείτε κυρία Κοκόνεν. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που ειναι μαλιστα εγω εψαχνα αλλου με συγχωρειτε κυρια κοκονεν αξιοτιμα μελη του κοινοβουλιου κυριε προεδρε σας ευχαριστω που καλεσατε την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στην ακρόαση αυτή. Και θα ήθελα καταρχήν να αναφερθώ και στην έκθεση την οποία εσείς συντάξατε και να σας εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για το ενδιαφέρον που δείχνει για το χώρο αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν μου δώσετε 10 λεπτά θα ήθελα να ξεκινήσω κάνοντας μία ε, παρουσίαση της δικής μας θέσης για τον πολιτισμό και το χώρο που έχει στην εξωτερική δράση και αν έχω χρόνο θα σας δώσω ένα-δύο παραδείγματα συγκεκριμένης δουλειάς που κάνουν οι αντιπροσωπείες μας στις τρίτες χώρες. Ο πολιτισμός παίζει ένα κομβικό ρόλο στο όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αναπτυξιακή εξωτερική πολιτική, έτσι ώστε να εξαλείψουμε την ε, φτώχεια και να πετύχουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο πολιτισμός αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο που μας βοηθά στο να ξεπεράσουμε τα προβλήματά μας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ενταχθεί σε όλες τις αναπτυξές και εξωτερικές πολιτικές που έχουμε και να καλέσουμε ε, όλα τα κράτη-μέλη να τοποθετήσουν τον πολιτισμό ε, σε θέση προτεραιότητας. Αυτές οι πολιτικές δράσεις ε, και κυρίως προς τις χώρες που βρίσκονται σε ανάπτυξη αποτελούν και βασικό πυλώνα της δικής μας δράσης. Και όταν λέω πολιτισμός, πιστεύω πως η προσέγγιση μας έχει ως στόχο να κάνει τον πολιτισμό ένα εργαλείο για την οικονομική και πολιτιστική και πολιτική πρόοδο, για τον εκδημοκρατισμό, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία έκφρασης. Και συγκεκριμένο παράδειγμα είναι το περιφερειακό μας πρόγραμμα στην ε, ε, νότια λεκάνη της ε, Μεσογείου με τα διάφορα οπτικοακουστικά προγράμματα που έχουμε χρηματοδοτήσει. Το όραμά μας για τον πολιτισμό ευθυγραμμίζεται με τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει σε διεθνές επίπεδο για να πετύχουμε τους στόχους ε, της σύμβασης της UNESCO που αποτελεί ένα αναπόσπαστο τμήμα του κοινοτικού κεκτημένου και βεβαίως αποτελεί και το βασικό πλαίσιο για την συνεργασία μας σε θέματα πολιτιστικά με τρίτες χώρες. Και από τότε που επικυρώθηκε η σύμβαση αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει δράση με στόχο να προωθήσει την επικύρωση σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι δράσεις αυτές έχουν να κάνουν με μια σειρά παρεμβάσεις, με πολιτική διαλόγου με τρίτες χώρες και διαπεριφερειακή συνεργασία, χρήση των υφιστάμενων και νέων εργαλείων και ad hoc δραστηριότητες που ευαισθητοποιούν ε, το κοινό για την ύπαρξη της σύμβασης. Και αυτή τη στιγμή ο ρυθμός επικύρωσης οδηγεί σε υψηλές προσδοκίες. Πιστεύουμε πως πολλοί ακόμα θα προχωρήσουν σε επικύρωση. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποίοι θα συνεχίσουν να προωθούν τη σύμβαση ως τον πυλώνα που αποτελεί την, το σημείο αναφοράς για την διακυβέρνηση των πολιτιστικών θεμάτων με τελικό στόχο ε, την σχεδόν καθολική ε, επικύρωση. Άρα και ισχύει. Για την εφαρμογή της σύμβασης είναι ε, στο, στην καρδιά της ατζέντα για τα πολιτιστικά θέματα και θα χρησιμοποιηθεί και με τη διάσταση της εξωτερικής πολιτικής. Έχουμε πολιτιστικό διάλογο με αρκετές τρίτες χώρες και είναι θέμα αρχής για την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει μία προχωρημένη θέση μέσω του διαλόγου για πολιστικά θέματα ε, και πολύ συχνά ζητάμε, από τους, πολύ συχνά καλούμε τους εταίρους μας στις τρίτες χώρες να επικυρώσουν τη σύμβαση αυτή. Ε, έχουμε λοιπόν ε, συνεχή διάλογο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Υπουργείων στην Ινδία, στην Κίνα, στο Μεξικό, στη Βραζιλία με ανταλλαγές που οδηγούν σε περαιτέρω εφαρμογή των όσων προωθούμε. Έχουμε και τις πολιτιστικές ρήτρες της Διεθνής συμφωνίες, ε, στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης, ε, στις συμφωνίες συνεργασίας αλλά και στα προγράμματα μακροπρόθεσμης στρατηγικής όπως επίσης και στα σχέδια δράση της διάφορες χώρες. Πιο συγκεκριμένα συνεργαζόμαστε με την UNESCO Έχουμε ένα πρωτόκολλο ε, συνεργασίας που ονομάζεται πολιτισμός και ε, χώρες που αναπτύσσονται. Είναι η πρώτη τεχνική παροχή βοήθειας που έχει ως σκοπό να ενισχύσει την ε, διαχείριση του πολιτισμού στις αναπτυσσόμενες χώρες και θα οδηγήσει στη μείωση της φτώχειας και στην ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, πώς το έχουμε στήσει όλο αυτό το εγχείρημα. Πριν την ακρόαση τηλεφώνησα στις αντιπροσωπείες μας, 137 αντιπροσωπείες έχουμε, και έλαβα μια εξαιρετική απάντηση. Έχω 50 παραδείγματα τα οποία θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Όπως έκανε και ο κύριος Διζανά, θα πω τι γίνεται στην Αίγυπτο. Η αντιπροσωπεία μας στην Αίγυπτο προσπαθεί να προωθήσει την ε, ε, πολιτιστική ποικιλομορφία και τις ε, και να προωθήσει τους πολιτιστικούς φορείς στη χώρα. Με προτάσεις οι οποίες έχουν προϋπολογισμό γύρω στα 200.000 ευρώ το χρόνο. Από το 2010 και μετά αυτή η πρόσκληση στην υποβολή προτάσεων έχουν επικεντρωθεί στη σύγχρονη τέχνη που δίνει πολλές ε, δυνατότητες για τον κοινωνικό και οικονομικό για την κοινωνική και οικονομική πρόοδο μιας χώρας. Και ίσως σας ενδιαφέρει να ξέρετε από τους δικαιούχους είναι πολιστικοί φορείς από τα κράτη-μέλη και ιδρύματα και για την Αίγυπτο Έχουμε το Ιταλικό Ινστιτούτο, την Ισπανική Πρεσβεία, το Ινστιτούτο Γκέτο, ε, το British Council και κάποιες ευρωπαϊκές πρεσβείες που έχουν συμμετάσχει. Κάποια καλά παραδείγματα είναι έργα που συνεργάζονται η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι δικαιούχες χώρες και τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη και ένα από αυτά ήταν το Φεστιβάλ Μεσογειακής Λογοτεχνίας το φεστιβάλ του ε, Κάιρο, ένα έργο με ντοκιμαντέρ για τα ανατέλλοντα αστέρια στην τέχνη. Όπως επίσης το πανόραμα ευρωπαϊκών ταινιών, κινηματογραφικών ταινιών, όπου συνεργάζονται οι πολιτιστικοί φορείς της ενδιαφερόμενης χώρας, των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εδώ πρέπει να τονίσω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει εφιστάμενες αιγυπτιακές δραστηριότητες και αυτό εξασφαλίζει την βιωσιμότητα αυτών των έργων. Έχουμε και κάποια άλλα που είναι μια, η δημιουργία μιας κοινή πλατφόρμας για τις πολιτικές, ευρωπαϊκές πολιτιστικές δραστηριότητες σε μια χώρα ε, που α, ε, κυρίως προωθεί τα πολιτιστικά έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει λοιπόν πάντα διάσταση της πολιτιστικής διπλωματίας και η συνεργασία μας προωθεί τους βασικούς, τις βασικές πολιτικές αξίες που χρειάζεται για την ανάπτυξη του πολιτιστικού κλάδου. Ελευθερία έκφρασης, δημιουργίας, προστασία και προώθηση της πολιτιστικής ε, ποικιλομορφίας και πρόσβαση στον πολιτισμό. Θα σταματήσω εδώ, θα μπορούσα να σας δώσω και πολύ περισσότερα παραδείγματα. Τι κάνει η αντιπροσωπεία μας στη Ρωσία. Κάνει καταπληκτικά πράγματα. Και με μεγάλη χαρά θα τα μοιραστώ μαζί σας αργότερα μπορώ να σας στείλω γραπτά. Να σας πω μόνο πως ήταν τόσο επιτυχής η, προ, η υποβολή ε, προτάσεων που πριν από μία ώρα μου έστειλαν μία πρόταση για πολιστικό έργο από το Γερεβάν της Αρμενίας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως πάντα θα έχει τελευταία το λόγο για να μας πει τη γνώμη σας και πρώτα θα μιλήσουν οι ε, ευρωβουλευτές και πρώτα η συνάδελφος. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που οργανώσατε την ακρόαση αυτή. Έρχεται την κατάλληλη στιγμή. Να ευχαριστήσω και τους ομιλητές για τα εισαγωγικά λόγια τα οποία είπαν. Στα πλαίσια της συνεργασίας με τους συναδέλφους για την έκθεση αυτή έλαβα πολλές πληροφορίες από διάφορους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, από διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι ουσιαστικά εντοπίζουμε τις ίδιε προτεραιότητες και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτή, από τη δική τους την πλευρά. Ορισμένε από τι προτεραιότητε αυτέ δεν είναι καινούριε. Επομένω, έχει έρθει η κατάλληλη στιγμή πλέον να περάσουμε από τα λόγια στην πράξη. Πρέπει να κάνουμε αυτό το επόμενο βήμα και πιστεύω ότι η δράση θα πρέπει να έρθει πλέον από την, το τομέα τη εξωτερική δράση, τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από το Συμβούλιο. Στι κάτω χώρε κάνουμε πολύ ποδήλατο. Και αν δεν συνεχίζει κανείς, αν δεν κουνάει κανείς τα πετάλια, πέφτει μετά από λίγο. Και φοβάμαι ότι αυτό συμβαίνει τελικά για με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τον πολιτισμό στην εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έκπληκτη βλέπω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Κοινωνία των Πολιτών, η Κίνα, το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένε Πολιτείε δίνουν μεγαλύτερη σημασία στο ζήτημα αυτό από ό,τι έχω δει εγώ σήμερα αλλά και στο παρελθόν στη συνεργασία που είχαμε με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση. Βλέπουμε ότι κάποια πράγματα γίνονται, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι υπάρχει ένας μεγάλος κατακαιρματισμός, ο οποίος ουσιαστικά λειτουργεί αρνητικά όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και τα απτά αποτελέσματα. Και αυτά βλέπουμε και στην πολιτική γειτονία. Πρώτον λοιπόν, το πρώτο με ερώτημα, τι πιστεύει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης όσον αφορά τη χρήση του πολιτισμού στα πλαίσια α, της οργάνωσης της θα μπει στον τομέα των επικοινωνιών, σε κάποιον άλλον τομέα δράσης της. Ποιες ευκαιρίες υπάρχουν ε, στα πλαίσια της χρησιμοποίησης του πολιτισμού για την δημοκρατική μετάβαση, για την εδραίωση της δημοκρατίας και ποια θα είναι η χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής γιατί βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση έχει εντοπίσει την πληροφορική ως σημαντική προτεραιότητα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά δεν ξέρω αν ε, στην πράξη θα δώσει όντως αυτή την ε, προσοχή. Θα μπορούσε ενδεχομένω να αναπτύξει περισσότερο το ζήτημα αυτό. Και μία ακόμα παρατήρηση. Σε μια εποχή οικονομικής ε, λιτότητας θα πρέπει να γνωρίσουμε ότι το hard power κοστίζει πολύ περισσότερο από ότι το να επενδύσουμε τελικά στον πολιτισμό, που θα μπορούσε να αποδώσει και πολύ περισσότερο στο μέλλον. Θα ήθελα λοιπόν να δω κάποια φιλόδοξα συγκεκριμένα σχέδια επί της ουσίας από αυτούς που εργάζονται στα πλαίσια της εξωτερικής πολιτικής. Ευχαριστώ Μαρέκη. Η κυρία Τρίπελ τώρα. Χάρη στους ε, ε, εμπειρογνώμονές μας θα ήθελα καταρχήν να μιλήσουμε ε, για τις ιδέες τις οποίες συζητάμε. Συζητάμε για την ήπια δύναμη, δηλαδή soft power. Ε, μιλάμε για κάτι που είναι και ήπιο και δυνατό. Ε, στην Κίνα υπάρχει η ε, ήπια δύναμη. Πιστεύω ότι εκεί υπάρχει περισσότερο στοιχείο της δυνάμεως. Υπάρχει και η ευρωπαϊκή λύση. Γι' αυτό χρειαζόμαστε περισσότερη σαφήνεια για το πώς εμείς ερμηνεύουμε την ήπια δύναμη για να καταλαβαίνουμε τι εννοούμε με το ήπιο και με το δυνατό. Και έρχομαι τώρα σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Ντουζαρντάν, ο οποίος ανέφερε ότι σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ιστορία η ήπια δύναμη απέβλεπε ε, στο να υποκινήσει το πνεύμα ανεκτικότητος στους ε, λαούς. Υπήρχαν λαοί οι οποίοι ήταν ε, αντίθετοι στην ισότητα και στην ανοχή, ε, και γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε όταν μιλάμε πόσο ορίζουμε ότι είναι δημοκρατικό, γενικό, με πνεύμα ισότητος, διότι διαφορετικά αν κοιτάξουμε τους πολέμους στα Βαλκάνια και την τρομοκρατία των Ναζί στη Γερμανία, πρέπει να ξέρουμε τι εννοούμε όταν μιλάμε για την δημοκρατική αρχή του πολιτισμού. Εάν λοιπόν καταλαβαίνουμε ποια είναι η ευρωπαϊκή προσέγγιση του soft power και αν θέλουμε να προωθήσουμε ειρηνικές επιλύσεις των διαμαχών δεν πρέπει να δίνουμε μαθήματα διότι ακόμη και αν κατανοούμε πλήρως τι είναι ο δημοκρατικός ο πολιτισμός ε, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε πολλές διαμάχες, πολλά προβλήματα με ε, την τρομοκρατία, με την, το σκεπτικό των Ναζί και δεν πρέπει να δίνουμε μαθήματα στις άλλες χώρες, πρέπει να δούμε τι είναι τα εσωτερικά μας προβλήματα και πώς μπορούμε να τα υπερβούμε για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε ε, σε πνεύμα ισοτιμίας χωρίς να δίνουμε μαθήματα στους άλλους. Και από δικιά μου άποψη θεωρώ ότι είναι πολύ βασικό ε, να έχουμε θεσμούς οι οποίοι προσπαθούν να συνεργαστούν και να έχουμε την ιδέα της νέας υπηρεσίας η οποία θα πρέπει καθημερινά να διεκπεραιώνει τέτοια θέματα και να εξηγούμε ε, γιατί ε, υπάρχει αυτή η ιδέα, αυτή η έννοια και ότι στα πλαίσια αυτά υπάρχει μία παρουσίαση για όσα θέλουμε να επιτύχουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φίσας, Σαντιάκο Φίσας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους εισηγητές γιατί νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπαν. Και να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ νομίζω πως για τον πολιτισμό δεν μας πιάνει κανείς. Η Ευρώπη είναι σε κρίση, σε κρίση οικονομική. Αλλά η δύναμη του ευρωπαϊκού πολιτισμού είναι κάτι το οποίο ξεπερνά αυτές τις δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες ζούμε και νομίζω ότι αυτό έχουμε καταφέρει και το έχουμε περάσει και στο εξωτερικό. Θα ήθελα να ρωτήσω κάποιους από τους εισηγητές ποια είναι η άποψή τους για τον συντονισμό που θα έπρεπε να υπάρχει μεταξύ αφενός αυτών των ιδρυμάτων που πολλά ε, ευρωπαϊκά κράτη έχουν στο εξωτερικό ε, και της ε, δουλειάς που κάνουν οι πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο εξωτερικό, γιατί πιστεύω πως οι πρέσβεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αντιπροσωπείες θα έπρεπε να προωθήσουν την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκού, του ευρωπαϊκού πολιτισμού, έτσι ώστε να κάνουν στο δυνατόν περισσότερο πολιτιστικές εκδηλώσεις για τα κράτη-μέλη εκεί που βρίσκονται. Και βέβαια, θα έπρεπε να δίνουν και πληροφορίες από πρώτο χέρι στους τοπικούς πληθυσμούς ε, που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη για να παραστούν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις σαν αυτά τα τεράστια φεστιβάλ που γίνονται ε, στις χώρες μας. Και νομίζω ότι αυτό και χρήμα θα φέρει και ο πολιτιστικός τουρισμός είναι μια ε, ελπίδα για το μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν η δράση μας να είναι ε, ε, κάτι το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη και που θα φέρει απτά αποτελέσματα. Ευχαριστώ λέει η πρόεδρος Σίλβια Κώστα. E Θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό και επίκαιρο διότι έχει σχέση με ε, τα θέματα που πραγματεύεται το Κοινοβούλιο σχετικά με τις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι όντως γεγονός ότι ε, ισχύει το θέμα αυτό του soft power, ε, ίσως όχι μονοθετικά αλλά και ιδιαίτερα στα πλαίσια των πολιτιστικών σχέσεων που προσπαθούν να νομιμοποιήσουν τις ε, πολιτικές ε, και διπλωματικές σχέσεις της Ευρώπης όπως το είπε και η συνάδελφος Τρούπελ δηλαδή υπάρχει ένα πνεύμα ηγεμονίας ευρωπαϊκής ή υπεροχής πολιτιστικής αλλά ελπίζω ότι μιλάμε για τις ίδιες αξίες και πιστεύω ότι υπάρχει, ε, υπάρχουν στοιχεία που ανέφεραν οι συνάδελφοι που κάθονται πίσω μου και που μπορεί να επιτρέψουν επιτρέψει στην Ευρώπη να μην υπάρχει μόνο μία παράλληλη ε, ε, εξέλιξη σαν αυτή η οποία υπάρχει στα κράτη-μέλη αλλά όπως ε, το είπε και η Πρόεδρος αυτή η διπλωματία μπορεί να αποτελέσει μία κρίσιμη μάζα η οποία θα επηρεάσει θετικά τις σχέσεις μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών. Μια κρίσιμη μάζα η οποία δεν θα εμπλέκεται υποχρεωτικά να πάσα στιγμή διότι πιστεύω ότι δεν πρέπει μόνο να εκφράζουμε ευχολόγια αλλά θα πρέπει να δώσουμε κάποιον προσανατολισμό. Τα κράτη-μέλη δεν πρέπει να εγκαταλείψουν την πολιτιστική τους ηγεμονία αλλά να συνεργαστούν διότι διαφορετικά η πολιτιστική πολιτική της Ευρώπης θα θεωρηθεί μόνο ένα παράλλη, μια παράλληλη πολιτική. Πρέπει να ενισχύσουμε δίκτυα στη Μεσόγειο, στη, το μεγάλο δίκτυο το οποίο υπάρχει ε, σχετικά με, τις, ε, με τα γεγονότα που ο δεν εκφράζονται παρκώς στην Ευρώπη την Ένωση Τηλεοράσεων με τρίτες χώρες που προσπαθούν να συσφίξουν τις σχέσεις τους στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ας παίξουμε λοιπόν τον ρόλο του καταλήτη και ας ενισχύσουμε την, ε, ε, το ρόλο αυτών των χωρών σε σχέση μαζί μας. Σκέφτομαι εδώ και της συνεργασίας. Και αναρωτιέμαι εάν θα μπορέσει να υπάρξει μία πιο συστηματική προσέγγιση από αυτές οι οποίες αναφέρθηκαν προηγουμένως κατά τρόπον ώστε οι ε, πολιτιστικές συνεργασίες να γίνουν πιο σαφείς. Υπάρχει και μία άλλη διάσταση στην συνθήκη της Λισαβόνας, το άρθρο 67 το οποίο ε, λέγει ότι πρέπει να ενισχύσουμε την ε, πολιτιστική διάσταση σε όλες τις πολιτικές κατά τρόπον ώστε να είναι πιο οριζόντιος. Θα έπρεπε λοιπόν να δούμε τις επιπτώσεις όλων των ευρωπαϊκών πολιτικών και συγχρόνως να υιοθετήσουμε μία προσέγγιση σεβόμενη την, ε, ε, τον πολιτισμό της ε, χώρας, πράγμα το οποίο θα εμπλουτίσει τις σχέσεις μας με αυτήν. Και πολύ σωστά το ανέφερε αυτό ο Γενικός Διευθυντής της Μποζάρ στις Βρυξέλλες. Το παράδειγμα το οποίο ανέφερε είναι ενδιαφέρον. και μπορούμε να αναπτύξουμε τα θέματα αυτά όχι μόνο στα κράτη-μέλη, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με ανάπτυξη πολιτικών και στρατηγικών κατά περιοχές, κατά ενότητες, ε, ε, όχι όλα τα θέματα μαζί, με μια πιο συνεκτική μέθοδο που θα αποβλέπει στην ενίσχυση των ε, διμερών σχέσεων. όχι απεικιοκρατικά αλλά με ε, αλληλεπίδραση. Έχουμε εξετάσει ε, πολιτιστικές ε, προτεραιότητες στην Ευρώπη παραδείγματος χάνην όπου συνεργαζόμαστε διότι αυτή είναι μία από τις εξωτερικές διαστάσεις Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ζητήσαμε να έχουμε έναν εκπρόσωπο και ε, θα έπρεπε να υπάρχει ο εκπρόσωπος αυτός σε όλες τις αντιπροσωπείες, δηλαδή όπου υπάρχει εξωτερική εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει ή όχι. Ευχαριστώ η κυρία Χάνιμπαλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πάντα θεωρούσα ότι ε, το ζήτημα αυτό ήταν αρκετά πολύπλοκο, όχι ιδιαίτερα εύκολο, γιατί είναι ιδιαίτερα γενικό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν του ομιλητέ που πιστεύω ότι μα βοήθησαν πολύ, τουλάχιστον εμένα με βοήθησαν να καταφέρω να καταλάβω κάπω καλύτερα το υποεξέταση ζήτημα. Αλλά από ό,τι φαίνεται μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Από τη μια μιλάμε για τη γενικότερη προώθηση του πολιτισμού και προσπαθούμε να δούμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση, τι κάνουν και άλλοι φορεί αν μπορεί να γίνει κάποια ανταλλαγή, ή συντονισμό προγραμμάτων και ήδη είχαμε κάποια θετικά παραδείγματα. Αλλά από την άλλη φαίνεται ότι μιλάμε και για ένα ευρύτερο ζήτημα. Δηλαδή πώ θα καταφέρουμε να οργανωθούμε στα πλαίσια της δημοκρατίας, πώς θα καταφέρουμε μέσω του πολιτισμού να προωθήσουμε την ειρηνική επίλυση των διενέξεων, Νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα δύο αυτά ζητήματα ως ξεχωριστά ζητήματα, μόλον ότι προσπαθούμε να τα εντάξουμε και τα δύο στα πλαίσια του πολιτισμού. Το ένα είναι καθαρά πολιτισμικό, ενώ το άλλο είναι περισσότερο πολιτικό, αν θέλετε, πολιτικός τρόπος για να ε, αναλαμβάνει κανείς δράση. Θα ήθελα λοιπόν να καταλήξουμε σε κάποιες πιο συγκεκριμένες συστάσεις, όπως είπε η κυρία Κώστα, μια κάποια στρατηγική, για να δούμε πώς θα καταφέρουμε να προωθήσουμε και τα δύο αυτά ζητήματα. Σαφώς θα πρέπει να βασιστούμε στα εφιστάμενα δίκτυα, αυτή είναι μια πολύ καλή ιδέα, δίκτυα τέτοια έχουμε παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ωστόσο, θα πρέπει να είμαστε και πολύ προσεκτικοί. Ένα ζήτημα το οποίο ήδη το θίξαμε, την πολιτιστική πολυμορφία. είναι πολύ εύκολο στα πλαίσια της πολιτισμικής συνεργασίας τελικά να ακούσουμε περισσότερα τα όσο να πούνε τα μεγάλα πολιτιστικά ιδρύματα και να ξεχάσουμε λίγο τα μικρά. Το Βρετανικό Συμβούλιο είναι παρόν παντού, μπορεί να επισκιάσει άλλους μικρούς οργανισμούς. Ας είμαστε προσεκτικοί ως προς αυτό λοιπόν και ας καταφέρουμε να φέρουμε με το μέρος μας στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής και κάποιες μικρότερες χώρες, οι οποίες μπορεί να μην έχουν ένα τόσο αναπτυγμένο δίκτυο πολιτιστικών Ινστιτούτων στα πλαίσια τώρα της προώθησης της πολιτικής αυτής κουλτούρας, της δημοκρατίας, της, α, της ειρηνικής διευθέτησης των διενέξεων, στα πλαίσια της πρόθεσης της λεγόμενης soft power της EPS δύναμης, Σίγουρα η ιδέα αυτή είναι πολύ σημαντική, είναι πολύτιμη, αλλά δύσκολα εφαρμόζεται στην πράξη. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με αυτό. Η συζήτηση όμω που έχει ήδη διεξαχθεί με βοήθησε πολύ να καταλάβω περισσότερο το ζήτημα. Κυρία Τάκολα. Κύριο Τάκολα, με συγχωρείτε. Yeah. Ε,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 Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ακούσαμε κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και από τους πρώτους εισηγητές που μας έκαναν την εισαγωγή αλλά και από τους συναδέλφους οι οποίοι αντέδρασαν στις προτάσεις αυτές. Και ακούσαμε και κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Νομίζω ότι όταν μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση το βασικό είναι να μιλάμε για μια κοινότητα αξιών. Δημοκρατία, ελευθερία έκφραση, οι αρχές οι δημοκρατικές και να ξεκινάμε από αυτή τη βάση. Είναι η κοινή πλατφόρμα, η βασική πλατφόρμα που αποτελεί αυτή την Ευρώπη με την πολλαπλή φωνή. Και νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε αυτές τις κοινέ αρχές τις οποίες όλοι μπορούμε να στηρίξουμε και επί των οποίων όλοι συμφωνούμε. Γιατί όταν κανείς ε, βλέπει τα πράγματα ε, από το εξωτερικό, ακόμα και σε πολιτιστικό επίπεδο, ε, μοιάζει η Ευρώπη να ακολουθεί διαφορετικά προγράμματα και ταχύτητες. Όταν λοιπόν σχολιάζουμε την ε, ψηφοφορία που έγινε πρόσφατα στην UNESCO για το θέμα της Παλαιστίνης και εκεί για μια φορά ακόμα η Ευρώπη δεν εκφράστηκε με μια ενιαία φωνή. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποια είναι τα κριτήρια τα οποία ακολουθούμε ε, και Πώ αντιμετωπίζουμε όλη την κοινή πολιτική μα κληρονομιά. Νομίζω πω θα πρέπει και στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση να, να έχουμε καλύτερη γνώση για το ποια είναι η πολιτιστική μα διαφορά. Για το να λέμε πω ε, στην περιοχή τη Μεσογείου ε, τα όσα συμβαίνουν συνδέονται με ε, το θρησκευτα, θρησκευτικά πιστεύω των λαών που ζουν εκεί δεν ε, αποτελεί την ιδανική ε, αντιμετώπιση των ε, καταστάσεων που αντιμετωπίζουμε για την Αραβική Άνοιξη, για παράδειγμα. Πρέπει να σας πω πως αποτελεί μια πρόκληση για την ε, περιοχή και σε πολιτιστικό επίπεδο. Πρέπει να δούμε ποια είναι η θέση του ατόμου μέσα σε κοινωνίες που έχουν διαφορετικές δομές από αυτές τις οποίες εμείς γνωρίζουμε. Άρα λοιπόν πρέπει να εξοικειωθούμε περισσότερο με την πολιτιστική πραγματικότητα και με τον τρόπο αυτό να προωθήσουμε το διάλογο. Εσείς είστε η τελευταία πριν από μένα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το ερώτημα το ακόλουθο θέλω να θέσω. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε μια πολιτιστική δημοπλατεία, διπλωματία η οποία θα περνάει κυρίως από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που ουσιαστικά θα περνάει κυρίως από τα κράτη-μέλη, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί από τις τρίτες χώρες με τις οποίες συνεργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ε, εμπλοκή στη δική του την ε, εσωτερική πολιτική. Επίσης, ε, θα θέλαμε να γνωρίζουμε πώς μπορούμε να έχουμε μία αποκεντρωμένη συνεργασία όσον αφορά την πολιτιστική προσέγγιση. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να παρέμβω. Καταρχήν είμαι πολύ ευτυχής ε, που είπε ο κύριος Βάγνερ ότι θα υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα αυτής της fact-finding mission, δηλαδή αυτής της αποστολής ε, ε, της αποστολής των αποτελεσμάτων και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να δούμε πώς ο δρόμος αυτός που ανοίξαμε θα ακολουθηθεί και θα προχωρήσει. Ε, πρέπει να ψάξουμε νέες δυνατότητες και να εμπλέξουμε και την κοινωνία των πολιτών. Μπορεί όμως να είναι και οι οργανώσεις ε, οι οποίες ε, όπως ελέγχθη τώρα είναι κρατικές οργανώσεις. Υπάρχουν όμως και άλλες οι οποίες ναι μεν χρηματοδοτούνται από το κράτος αλλά δεν θεωρώ ότι το Ινστιτούτο Γκέτε το διευθύνει η κυρία Μέρκελε που δεν είναι λόγο και υποθέτω ότι και σε άλλες χώρες συμβαίνουν παρεμφερή γεγονότα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε τη δυνατότητα να εμπλέξουμε επιτόπου την κοινωνία των πολιτών. Γι' αυτό και χαίρομαι που είπαν διάφοροι ε, σχετικά με την Αραβική Άνοιξη ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερο όσον αφορά την υποδομή αλλά θα πρέπει να προωθήσουμε και την δημοκρατία πρέπει να, τη, να στηρίξουμε τις ενέργειες αυτές με πολιτιστικές και πολύ σωστά είπε η κυρία Τρίπελ, βέβαια δεν θα πάμε εκεί άοπλοι, ε, όλοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητές μας, να επωφεληθούμε. Και δεν μιλάω μόνο για την Αφρική αλλά και για την Ασία, την Κίνα, την Αμερική. Παντού πρέπει να διηγηθούμε την ευρωπαϊκή μας ιστορία δηλαδή αυτό που είπε ο κύριος Φέντερ, ε, αυτό το οποίο πρέπει να προωθήσουμε και που καταναλώνουμε και γι' αυτό χρειαζόμαστε και την ταινία. Όχι μόνο τα ντοκιμοντέρ αλλά και γενικώ ταινίε διότι εκεί εξηγούμε και διηγούμαστε τις ευρωπαϊκές μας ιστορίες και υπάρχει ένα μια μεγάλη έκθεση, η ντέφα του συναδέλφου Μπίσκι. Ε, θα πρέπει λοιπόν να ενδιαφερόμαστε και τότε θα πρέπει να μπορέσουμε να το μεταδώσουμε και προς τα έξω και γι' αυτό χαίρομαι ότι οι δύο Γερμανοί που κέρδισαν το βραβείο Λούξ προπέντε τόν και πέρυσι ε, μεταφράστηκαν σε άλλες γλώσσες ε, νομίζω ότι ε, πέραν των γλωσσών που μεταφράστηκαν επισήμως συνέβαλε με άλλες εννέα γλώσσες και το Ινστιτούτο Γκέτε θα μπορέσουμε μπορέσουμε λοιπόν τώρα να βρούμε ε, έναν ομόλογο του Γκέτε σε μια άλλη χώρα. Παραδείγματο χάρη στη Γαλλία με το Institut Français ε, για μια βελγική ταινία η οποία θα πρέπει να προβληθεί στην Ασία, στην Αμερική για να μπορέσουμε να προωθήσουμε πολιτιστικά θέματα και ε, να αντεπεξέλθουμε των ε, δυσχεριών Πρέπει δηλαδή να έχουμε τρόπο να προωθήσουμε την πολιτιστική μας πολυμορφία. Μετά, όσον αφορά τον υπεύθυνο η το, την πρεσβεία, θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένος, πρέπει να ασχολείται μόνο με τον πολιτισμό. Χρειαζόμαστε εις τα, στις ευρωπαϊκές πρεσβείες κάποιον που θα αναλάβει αυτά τα θέματα και θα μπορέσει να να βοηθήσει, να, μας πει πώς αυτό θα προχωρήσει. Διότι γενικώ χρειαζόμαστε ε, ένα άτομο το οποίο θα είναι κατηρτισμένο πολιτιστικά αλλά μήπως χρειαστεί και περαιτέρω επιμόρφωση ε, ε, παραδείγματος χάρη ε, ένα γραφείο το οποίο θα προσπαθήσει σε κάθε ευρωπαϊκή εκπροσώπηση να υπάρχει ένα τέτοιο άτομο και δεν σημαίνει ότι όποιος είναι Άγγλος θα ασχοληθεί με τα Αγγλικά και ο Γάλλος με τα Γαλλικά αλλά θα προσπαθήσει να φέρει σε επαφή τους τοπικούς παράγοντες με τους ευρωπαϊκούς ε, νομίζω ότι σήμερα ελέγχθησαν εδώ ενδιαφέροντα πράγματα και ελπίζω ότι κατόπιν αυτών τα οποία συζητήσαμε μπορούμε να κλείσουμε. Νομίζω δε ότι η Κατερίνα το ανέφερε αυτό και πέραν αυτού θα πρέπει να συμπεριληφθεί και άλλο στοιχείο πέραν του πολιτισμού. Δηλαδή θα πρέπει να εμπλέξουμε όλους αυτούς που το επιθυμούν, όσους εργάζονται στις διάφορες επιτροπές. Και όταν μιλάμε για την εξωτερική υπηρεσία θα πρέπει να εμπλέξουμε και τις εξωτερικές σχέσεις και το εξωτερικό εμπόριο. Θα υπάρχει επιπρόσθετη χρηματοδότηση και θα ευαισθητοποιηθούν για τις μεγάλες δυνατότητες οι οποίες προσφέρονται για να εμπλακούμε όλοι. Καλό θα ήταν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι αυτό ελέγχθη εμέσως ε, ε, μπορέσουν να διευρυνθούν οι ε, έδρες ζωμονέ ε, παραδείγματος χάρη ε, στο Πανεπιστήμιο του Καΐρου, στο Τορόντο ή οπουδήποτε διότι ενδεχομένως έχει γίνει αλλά ναι πέστε το και στην κυρία Κοκόνεν <coughs> ή δεν θυμάμαι ποιος άλλος ήταν είπατε ότι πρέπει να μιλάμε περισσότερο και να διδάσκουμε περισσότερο για την Ευρώπη. Αλλά το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το οποίο μας προσφέρατε και μας είπατε να κάνουμε προς τα έξω θα πρέπει καταρχήν να γίνει εδώ. Για πηγαίνετε στα σχολεία μας, για δέστε ότι δεν μιλάμε για την Ευρώπη στα σχολεία όπως θα έπρεπε. Άρα αυτό που προτείνουμε είναι πρώτα πρώτα να ασχοληθούμε με τα του οίκου μας και μετά άπαξ και θα έχουμε αποκρισταλωμένες ιδέες να τις προωθήσουμε προς τα έξω. Και τώρα δίνω το λόγο ο καθένας από τους παρεμβαίνοντες για πέντε λεπτά και μετά η Επιτροπή θα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση αυτή. Σε τρεις σημεία θα ήθελα να επιμείνω. Πρώτον, όντως ο πολιτισμός δεν είναι μια αθώα λέξη και πολλές διενέξεις, πολλοί πόλεμοι ουσιαστικά χρησιμοποιούν, έχουν ε, κάποιους κάποιες πολιτισμικές αιτίες ή χρησιμοποιούνται πολιτισμικά. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα πρέπει να δώσουμε στρατηγική σημασία στη χρήση του πολιτισμού στο μέλλον. Πρόσφατα δίδασκα για, τα, για την πολιτισμική διπλωματία, για την έννοια της ήπιας δύναμης και Κοιτούσα έξω από το παράθυρο της αίθουσας στην οποία βρισκόμουν και έβλεπα ένα κτίριο το οποίο ήταν ακόμα κατεστραμμένο μετά τους βομβαρδισμούς του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να γνωρίζουμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ήπια αυτή δύναμη. Και στο παρελθόν γνωρίζαμε τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει. Η Ακαδημία των Επιστημών είχε την απαραίτητη γνώση, αλλά παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κατάφερε να ασχοληθεί σοβαρά με τα πολιτισμικά αυτά εργαλεία. Τα έχουμε πλέον αυτά στα χέρια μας, επομένως ε, στο μέλλον δεν χρειαζόμαστε απλώς τις βέλτιστες πρακτικές. Οι βέλτιστες πρακτικές αποτελούν τη βάση για το παν και χαίρομαι πάρα πολύ που η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης προσπαθεί να συλλέξει σε επίπεδο αντιπροσωπιών όλη αυτή την εμπειρία βέλτιστων πρακτικών. Θα πρέπει όμως να γνωρίσουμε και πάνω σε ποιες άλλες ευρωπαϊκές θεμελιώδεις αξίες μπορούμε να βασιστούμε. Τι μπορούμε να συζητήσουμε εσωτερικά και εξωτερικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς μπορούμε να αποφύγουμε την υποκρισία πώς θα καταφέρουμε να προστατεύσουμε αυτή την αυτοκρατική μας που είναι μέρος της ευρωπαϊκής πολιτισμικής κληρονομιάς. Και κάτι ακόμα. Η στρατηγική αυτή και πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί στο μέλλον. Η στρατηγική αυτή δεν έχει να κάνει βέβαια με την δημιουργία τεράστιων έργων, οδικών υποδομών ή ενεργειακών υποδομών. Χρειαζόμαστε στα πλαίσια του πολιτισμού πολλά διαφορετικά μέσα και όχι ένα και μοναδικό μέσο. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας διαθεσμικός διάλογος, ο οποίος θα καταλήξει στα κατάλληλα μέσα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον πολιτισμό, ιδίω απέναντι στις τρεις χώρες. Για παράδειγμα, Γνωρίζω δύο συναδέλφους από την ε, Λευκορωσία. Ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προσπαθήσει να κάνει σπουδαία πράγματα στη χώρα αυτή, αλλά ουσιαστικά δεν κατάφερε να ελοποιήσει τις αρχικές της ιδέες. Έχω μιλήσει με δύο καλλιτέχνες από την χώρα αυτή, που μου είπαν ότι τελικά δεν κατάφεραν να αποφεληθούν από την ε, κοινοτική υποστήριξη. Κριτική μάζα τέλος. Συμφωνώ ότι στη συνεργασία που θα πρέπει να έχουμε ανάμεσα στην κοινωνία των πολιτών, τους πολιτικούς ηθήνοντες, τους κρατικούς ηθήνοντες. Σαφώς θα πρέπει να δημιουργηθεί μια κριτική μάζα στη συνεργασία αυτή. Είναι όμως σημαντικό να γνωρίζουμε το ακόλουθο, αν οι εθνικά ενδιαφερόμενοι μόνο αυτοί οι οποίοι θα συνεργαστούν μεταξύ του, θα είναι δύσκολο να πετύχουμε ένα ευρωπαϊκό αποτέλεσμα. Τα εθνικά αυτά δίκτυα, οι εθνικοί οργανισμοί, οι οργανισμοί είναι σαφώ η βάση, θα πρέπει να του προστατεύσουμε, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και κάποια ευρωπαϊκή συνιστόσα στη στρατηγική. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο πιστεύω ότι ε, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση ε, θα πρέπει ε, να δει πω μπορεί να ανταποκριθεί στο ζήτημα αυτό και από πολιτική πλευρά Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Κατρίνκα. Να ξεκινήσω λοιπόν και εγώ το, με το τι σημαίνει αυτή η χαλαρή δύναμη, το soft power. Όταν κανείς μιλά για την Κίνα και εκεί μιλάμε για 300 ιδρύματα πολιστικά, δεν νομίζω ότι πρόκειται για χαλαρή δύναμη, νομίζω πρόκειται για πολιτιστική εξαγωγή. Και εμείς δεν θα κάνουμε κάτι αντίστοιχο, δεν θα εξάγουμε πολιτισμό και τέχνης. Πολύ μεγάλη διαφορά για το τι κάνουμε στο εσωτερικό προσπαθώντας να καταλάβουμε το ιστορικό υπόβαθρο όλων των κρατομέλων, την ε, παραδοσιακή τους δημιουργική έκφραση, τις γλώσσες, όλα αυτά προσπαθούμε να τα ε, εξηγήσουμε στον εξωτερικό κόσμο και να προχωρήσουμε σε διάλογο. Και όχι μόνο προς την Κίνα και προς τις Ηνωμένε Πολιτείες, για παράδειγμα, γιατί ξέρω πολύ καλά αυτά τα ιδρύματα και πρέπει να σου πω ότι εξάγουν. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά από την Ευρώπη και πρέπει να το δεχτούμε και να το χωνέψουμε. Πολύ σωστά. Έχουμε πάρα πολλά θέματα τα οποία είναι πανευρωπαϊκά, πανευρωπαϊκής σημασίας, για παράδειγμα τη μετανάστευση, τις σειράξεις, ή κάτι που είναι πιο ουδέτερο, αλλά μπορεί να είναι εξίσου ακα... την πολυγλωσία. Όλα αυτά τα θέματα λοιπόν αντιμετωπίζονται και έχουμε συλλέξει πάρα πολλά παραδείγματα σε χώρες που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα, για παράδειγμα όπως στην Αφρική. Ακόμα αυτό το σχέδιο βρίσκεται σε εξέλιξη. Και δεν είναι μόνο τις δικές μας ιστορίες, όχι. Ακούμε και τα όσα μας αφηγούνται από το εξωτερικό. Και καλούμε στις χώρες μας, δεν πηγαίνουμε μόνο. Για μένα λοιπόν αυτά είναι πολύ σημαντικά. Και βέβαια εδώ αυτό άπτεται ε, της κινητικότητας το θέμα, γιατί είπαμε προς τα έξω αλλά και προς το εσωτερικό. Το δεύτερο που είναι ίσως και πιο πρακτικής φύσης είναι η οργάνωση και η διαχείριση αυτών. Πείτε μου, πού μπορεί να φτάσει κανείς. Γιατί εγώ είμαι πολύ ρεαλίστρια και γι' αυτό κάνω πάντα αυτή την ερώτηση. Έχετε κάποια σχέδια εσείς, έχετε ανθρώπους με συγκεκριμένε αρμοδιότητες, θα εκπαιδεύσετε προσωπικό για τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι σημαντικό. Εγώ ξέρω πολλούς που ξέρουν πολλά. Αλλά ο περισσότερος κόσμος δεν καταλαβαίνει πως ο ευρωπαϊκός πολιτισμός αποτελείται από ε, μία συλλογή των τοπικών εθνικών πολιτισμών. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει ένας ενιαίος πανευρωπαϊκός πολιτισμός. Και οι περισσότερες αντιπροσωπείες δεν φταίνε, αλλά είναι αρκετά αθώες στο χώρο αυτό και ίσως θα έπρεπε να εκπαιδευτούν καλύτερα. Κατρίνκα κλείσε το μικρόφωνο σου και τώρα ο κύριος Ντουζαντά. Θαυμάσιο όνομα. Ευχαριστώ. Ναι, είχαμε πώληση ενδυμάτων παιδικών σχετικά με το soft power. Θα ήθελα να πω ότι δεν μπόρεσα στο χρόνο μου να το αναπτύξω, αλλά ίσως η Ευρώπη μετά από πάρα πολλά χρόνια θρησκευτικών πολέμων μεταξύ καθολικών και διαμαρτυρωμένων ε, διαπίστωσε τι μπορούσε να αποτελέσει ε, μία πρόοδο και γι' αυτό πιστεύω ότι σχετικά με τον Μποζάρ όλοι συμφωνούμε για αυτή την προοπτική της Ευρώπης αλλά προσωπικά πιστεύω βάσει του ποιες ήταν οι ε, απαντήσεις σήμερα δεν υπάρχει κανείς που μπορεί να κάνει σωστά αυτή τη δουλειά και αυτό εξαρτάται από την καλή θέληση των ε, πρέσβεων ε, και ελπίζουμε ότι οι διμερείς ε, Ευρωπαίοι ε, πρέσβεις θα μπορέσουν να αναλάβουν αυτό το έργο σε ολόκληρο τον κόσμο και φοβάμαι κάπως ότι αν μιλήσουμε για τον Πίτερ Κόμες και τι έγινε στην Ισπανία το περασμένη Κυριακή δεν θα έχουν πλέον Υπουργό Πολιτισμού στην Ισπανία και θέλουν να συγχωνεύσουν ε, το Υπουργείο Οικονομίας, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Πολιτισμού ε, με το Ινστιτούτο ε, Θερβάντες και άλλα, όλα αυτά να συγχωνευτούν και μακροπρόθεσμα μπορεί να υπάρχει προ, προ, βλήμα κρίσιμης μάζας. Όσον αφορά την ε, Κίνα, υπάρχει μεν εκεί ε, μία κατάσταση, αλλά μην ξεχνάμε και άλλες περιοχές όπως οι χώρες BRIC και υπάρχουν και ευρωπαϊκές ε, αναπτυσσόμενες χώρες γιατί μιλάμε για χώρες οι οποίες είναι σημαντικές και έγινε εδώ μία διάσκεψη κορυφής ε, στις Βρυξέλλες υπό τον Επίτροπο Μισελ ε, μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής. Ε, δεν πρέπει λοιπόν να ξεχνάμε όταν μιλάμε για την Ινδία και για την Κίνα τις άλλες χώρες και σας υπενθυμίζω ότι η γενική εκπρόσωπος εις την Ευρωπαϊκή Ένωση μάλωσε τους υπευθύνους ότι ε, δεν προωθούνται επικοδομητικά οι πολιτιστικές σχέσεις. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Ε, υπάρχουν ε, οι επιθυμίες των Κινέζων, των Ινδών και άλλων να συνεργαστούν με την Ευρώπη και όχι μόνο εμπορικά ή οικονομικά γιατί είχα κληθεί στις Ηνωμένε Πολιτείε και θυμάμαι ότι στη δεκαετία του 70 και του 80 δεν υπάρχει πλέον υπηρεσία για τον πολιτισμό έχουν επικεντρωθεί στην Αφρική ε, και με είχε καλέσει τότε μια αμερικανική ε, υπηρεσία για λόγους προπαγάνδας. Μπορούμε λοιπόν να προωθήσουμε προγράμματα και αν κάνουμε κοινά προγράμματα με τους ε, Ινδούς και με τους Κινέζους θα πρέπει να είναι εξαιρετικά. Δηλαδή <clears throat> όταν πήγαμε ή στο Πεκίνο χρειάστηκε να συνεργαστούμε με τους υπευθύνους και ε, ε, για ε, να κάνουμε εδώ το αντίστοιχο πρόγραμμα επιτύχαμε να περιληφθούν εδώ θέματα που δεν μπορούσαν να παρουσιαστούν στην πλατεία Τιέναν Μεν και αυτό συμβαίνει και σε άλλες χώρες με ε, ε, ε, άλλα, ιδρύματα όπως το Ινστιτούτο du Monde και άλλα. Αλλά το Ινστιτούτο Γιουμπερκιάν, το Ινστιτούτο du Monde ή άλλα έχουν στραφεί προς διμερείς σχέσεις τα τελευταία χρόνια. Και αν κοιτάξετε τη το γεωπολιτικό χώρο πρέπει να είμαστε πιο συστηματικοί και γι' αυτό στο Μποζάρ ζητάμε να καταρτιστεί μία πολυμερής πλατφόρμα σχέσεων και, μικρή και μικρά και μεγάλα ιδρύματα να συμμετάσχουν όχι για λόγους προπαγάνδας, προσπαθούμε να είμαστε ανεξάρτητοι σε όλα αυτά τα θέματα, και αναφέρομαι εδώ τώρα στην έδρα Ζωμονέ παραδείγματος χάρη του Καΐρου ε, αλλά σήμερα στο Κάιρο ε, δεν υπάρχει μεν ε, έδρα Ζωμονέ υπάρχει όμως Αμερικανικό Πανεπιστήμιο και ενώ δεν υπάρχει Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Ελπίζω λοιπόν ότι θα έχουμε μεγαλύτερες φιλοδοξίες και, και αύριο θα μπορέσουμε να συνδυάσουμε την παιδεία με τον πολιτισμό και αυτές οι διασυνδέσεις σε πολυμερής συνεργασίας μεταξύ διαφόρων επιτρόπων, ο κύριος Φίλε παραδείγματος χάρη με άλλους συναδέλφους που θα συμμετάσχουν σε αυτές τις συζητήσεις. Θα είχα να πω κι άλλα, αλλά εδώ έχετε ένα γενικό πλαίσιο. Η κυρία Φιλικάινεν. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά την έννοια του soft power της ήπιας δύναμης, θα αναφερθώ σύντομα σε αυτό. Η συζήτηση είναι πολύ σημαντική, επομένως θα πρέπει να αναφερθούμε λίγο περισσότερο σε αυτόν τον ορισμό. Υπάρχει μία έννοια του soft power, μία και μοναδική, αλλά πολύ διαφορετική τρόπη μπορεί κανείς να υλοποιήσει το soft power. Άλλο είναι ο τρόπο με τον οποίο υλοποιεί το soft power η Κίνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική όταν προσπαθεί να ασκήσει την δική τη soft power, η δύναμη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα άλλο προτέρημα, ένα άλλο προνόμιο. Έχει μια δημοκρατική προσέγγιση, μια δημοκρατική παράδοση. Οτιδήποτε και να αποφασίσει να προωθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον θα έχει την υποστήριξη ενός δημοκρατικού κοινού, θα υπάρχει μια δημοκρατική βάση. Επίσης, κατά την άποψή μου, το soft power έχει ένα ακόμα προνόμενο και μειονέκτημα. Είναι μια έννοια πολύ ανοιχτή στον διάλογο, αν τη συγκρίνουμε με άλλες μορφές άσκησης εξουσίας. Από την άλλη όμως, η ήπια δύναμη πολλές φορές δεν γίνεται τόσο ορατή, το αντίθετο μάλιστα. Με αποτέλεσμα να απαιτείται μια πολύ πιο ε, προσεκτική προσέγγιση προκειμένου να καταφέρουμε να εντοπίσουμε την δράση του soft power. Χαίρομαι πάρα πολύ πάντως που η έκθεσή σας αναφέρεται στο ζήτημα αυτό. Όσον αφορά τώρα το ευρωπαϊκό μοντέλο στο οποίο αναφέρθηκα, ιδίως όταν ε, πήρα τον λόγο για να πω ότι θα πρέπει σε αυτό να επικεντρωθεί το soft power της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της πολιτισμικής διπλωματίας θα μπορέσει να διαχύσει περισσότερο τις θετικές εμπειρίες που έχει για την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων. Θα καταφέρει να προωθήσει το μοναδικό πολιτικό και δικαστικό της σύστημα σε παγκόσμιο επίπεδο υφίσταται μια τέτοια ανάγκη και πολλές φορές βλέπουμε ότι σε διεθνές επίπεδο ή σε περιφερειακό επίπεδο θα μπορούσαν να υπάρξουν τέτοιες ανταλλαγές στις οποίες θα μπορούσε να συμβάλλει πολύ με την εμπειρία της Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσε λοιπόν σε αυτό το πολιτικό πλαίσιο να δραστηριοποιηθεί η πολιτισμική διπλωματία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος για μισό λεπτό ήθελε να πει κάτι αλλά για μισό λεπτό, πολύ σύντομα παρακαλώ. Ήθελα να πω το εξή Η συζήτηση που διεξάγεται εδώ και η πηγή πληροφοριών είναι ο Φρεντερίκ. Είναι μια συζήτηση που γίνεται από τεχνοκράτες. Θα πρέπει λοιπόν κάποιοι καλλιτέχνες, κάποιοι δημιουργοί να μπουν στη συζήτηση. Ξέρω πως ε, στις 8 Δεκεμβρίου το λόμπι που θα έρθει στο Μποζάρ θα φέρει και κάποιους καλλιτέχνες, αλλά νομίζω ότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τη θέση των δημιουργών και καλλιτεχνών στο μέλλον στη συζήτηση αυτή. Κυρία Κοκόνεν, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πάρα πολλά θέματα, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, να ξεκινήσω με το θέμα της ε, ε, του προσωπικού που έθεσε στην έκθεση ο κύριος και στη δημιουργία διευθύνσεων. Κοιτάξτε, οι δημοσιονομικοί περιορισμοί είναι τέτοιοι που μόνο ο συντονισμός και η ομαδοποίηση των πόρων επιτρέπονται. Και αν αναρωτιόσαστε γιατί κάποιος ήρθε σήμερα, κάποιος από τη δική μου διεύθυνση να μιλήσει για τον πολιτισμό, σας είπα ότι εγώ συντονίζω αυτή τη στιγμή με τις αντιπροσωπίες για να έχω μια εικόνα του τι γίνεται επί τόπου και εμείς συντονίζουμε από, τη δική μου, από το δικό μου τμήμα. Κατευθύνουμε, βοηθάμε, συνδράμουμε. Αλλά το είπα και στην αρχή της παρουσίασής μου. Η πολιτική διάσταση βρίσκεται στον πυρήνα και αποτελεί προτεραιότητα όλων των αναπτυξιακών πολιτικών. Άρα λοιπόν γίνεται κάποιο mainstreaming. Αυτός ο συντονισμός δεν είναι μόνο η στρατηγική επικοινωνία που συντονίζεται με τις αντιπροσωπείες, αλλά και οι αντιπροσωπείες συντονίζονται μεταξύ τους επί τόπου. Πολύ συχνά ε, έρχονται οι πολιτιστικοί ε, ε, ατασέ και συνεδριάζουν. Και για τη Ρωσία, εκτός από τα κοινά project ε, συζητάνε μεταξύ τους το τι γίνεται με τα πολιτιστικά ιδρύματα στη Ρωσία σχέση με τις αρχές της ρωσικές ε, βίζες για ε, τους Ευρωπαίους καλλιτέχνες, εισαγωγή μουσικών οργάνων για τις συναυλίες, αυτά. Είναι λίγα από αυτά που κάνουν. Θεσμικά εμείς συντονίζουμε μέσω της δικής μας επιτροπής μέσω του δικού μου τμήματο που είναι η Επιτροπή Στρατηγικής επικοινωνία, και κάνουμε συνεδριάσεις ε, στην Επιτροπή την αρμόδια, η οποία πολύ ε, σύντομα θα συνεδριάσει και για θέματα πολιτισμού και θα σας καλέσουμε. Η ερώτηση κυρία Σάρκια για το ποια είναι η άποψή μας για τον πολιτισμό η πολιτική διπλωματία αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της δικής μας διπλωματίας. Η πολιτική διπλωματία, η ψηφιακή διπλωματία. Άρα λοιπόν συνεργαζόμαστε και με τις ε, σχετικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια της αρμόδιας επιτροπής που ε, προανέφερα. Τώρα για το, τις προσλήψεις στις αντιπροσωπείες όπου ζητήσατε να έχουμε κάποιον σύμβουλο για πολιτικά θέματα ε, ή πολιτιστικό επιτετραμένο για παράδειγμα, να σας πω πως έχουμε μικρές αντιπροσωπείς όπως στην ε, ε, Βολιβία. Έχουμε μία τεράστια στην Ουάσιγκτον που έχει τέτοια θέση. Η πραγματικότητα είναι πως στις μικρές αντιπροσωπείες οι αξιωματούχοι για θέματα τύπου και ενημέρωσης μπορεί να συντονίζουν και τα θέματα τα πολιτιστικά. θα χαρείτε για την ταινία ε, γιατί τώρα που κάνουμε την απογραφή με το τι κάνουν οι αντιπροσωπείες 50 αντιπροσωπείες απάντησαν και 37 ε, μας είπαν πως οργανώνουν πολύ μεγάλα φεστιβάλ Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου. Άρα λοιπόν γίνεται προώθηση του Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου σε τρίτες χώρες. Για τα δίκτυα θα σας αφήσω αυτό τον πίνακα έχω η αντίτυπα και όταν το διαβάσετε θα δείτε πως πολλές από τις αντιπροσωπείες συνεργάζονται με τα τοπικά ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, όπως επίσης και με τη Γιούνις. Οπότε η, η δουλειά γίνεται και χαίρομαι που μπορώ να σας το αναφέρω. Ευχαριστώ, θα σας ξανακαλέσουμε. Και τώρα θέλω να δώσω το λόγο στον Ισπανό συνάδελφο για να μπορέσει να απαντήσει στον κύριο Ντουζαντά. Αλλά παρακαλώ γρήγορα, δεν έχει ακόμη κυβέρνηση. Εγώ δεν ξέρω τι θα κάνει ο Μαριάνο Ραχώη που θα είναι ο νέος Πρωθυπουργό, Αλλά από τις πληροφορίες που έχω και από τα όσα διάβασα στον τύπο, όντως θα γίνει Γενική Διεύθυνση το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτό είχε γίνει και υπό την Πρωθυπουργία του κ. Ασνάρ γιατί στην Ισπανία οι αρμοδιότητες του πολιτισμού ανήκουν ε, στις, αυτόνομες, στις αυτονομίες. Ε, το η κεντρική κυβέρνηση έχει λίγες πολιτικές αρμοδιότητες. Οπότε έχοντας μια γενική γραμματεία η οποία θα ανήκει στο Πρωθυπουργικό Γραφείο θα εξυπηρετήσουμε δύο στόχους. Πρώτα απ' όλα να δημιουργήσουμε αυτή την, το νέο νόμο για τις χορηγίες και δεύτερον εξωτερική προώθηση ε, του πολιτισμού και της ισπανικής γλώσσας. Γιατί μέχρι τώρα τα Ινστιτούτα Θερβάντες ε, ε, ήταν τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών, θα περάσουν τώρα στη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού και θα φύγουν από το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων. Λοιπόν, ο καθένας έχει τα δικά του. Και αν δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει κύριε Ντουζαρντάν δεν θα πρέπει να βρίζουμε. Να είμαστε αισιόδοξοι και να ελπίσουμε ότι η Ισπανία είναι μια πολιτιστική χώρα η οποία δεν θα μείνει πίσω. Λοιπόν, τώρα η εκπρόσωπος της Πολωνικής Προεδρίας έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την ε, εκδήλωση και τη θαυμάσια ευκαιρία που μου δώσατε να συμμετάσχω σε αυτή τη συζήτηση. Όπως ελέγχθη, στο σημερινό κόσμο υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα, αλλαγές στις επικοινωνίες και αυτό προωθεί τη σημασία της soft power, της υπείας δυνάμεως όπως την ε, αναφέραμε. Ε, οι ανταλλαγές, ο διάλογος ε, είναι κάτι το οποίο υπάρχει σε γενική σε γενικό πλαίσιο αλλά επίσης εις τον τομέα της προωθήσεως και υπάρχει ε, μία δυνατότητα μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητος. Οπότε αυτός ο τρόπος του σκέπτεστε θα πρέπει να προωθηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μία συζήτηση σαν τη σημερινή ε, δεν είναι μοναδική. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα θέματα αυτά ενδιαφέρουν ε, ιδιαίτερο την Επιτροπή Πολιτισμού και μετά από το 2007 όπου το Συμβούλιο υιοθέτησε το πρόγραμμα προωθήσεως των πολιτιστικών εκδηλώσεων αποτελεί ο τομέας αυτός ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έχουμε μακροπρόθεσμα προγράμματα εργασίας του Συμβουλίου για τα μέτρα αυτά και τα έχουμε υιοθετήσει όσον αφορά το πρόγραμμα εργασίας 2008-2010 είχαμε προωθήσει ε, την ε, ε, συμφωνία της UNESCO για τις μορφές εκφράσεως δεν περιοριστήκαμε όμως μόνο σε αυτά το 2008 είχαμε <clears throat> περιλάβει στα συμπεράσματα του Συμβουλίου την πολιτιστική πολυμορφία και τον πολιτιστικό διάλογο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των κρατών μελών. Και, και όσον αφορά τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, κινήσαμε το ενδιαφέρον. Όσον αφορά το πρόγραμμα μέχρι το 2014 προβλέπονται συγκεκριμένα μέτρα για την πρόθεση του πολιτισμού Μία πρώτη συνάντηση επετεύχθη κατά την Ουγγρική Προεδρία στο ΠΕΤΣ φέτος τον Ιούνιο και αναφερθήκαμε στη συνολική, περιφερειακή και τοπική προοπτική. Και η Πολωνική Προεδρία στο Λουμπλίν οργάνωσε μία παρεμφερή συνάντηση κατά τρόπον ώστε να υπάρξουν ε, ε, διπλωματικές ανταλλαγές ιδίως στα πλαίσια των πολιτιστικών ανταλλαγών και δεν συμμετείχαν μόνο δημόσιοι υπάλληλοι των ευρωπαϊκών χωρών αλλά και εκπρόσωποι των επιστημών όπως άλλωστε και εκπρόσωποι ε, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, ήταν η κυρία Μαρία Κοκόνεν σαν εκπρόσωπος ε, της Γενικής Διευθύνσεως και από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης η κυρία Λαϊτίνεν. Ε, επιπλέον ε, ε, είχαμε μία βιντεοδιάσκεψη με την κυρία Σάκε Ευρωβουλευτίνα στην οποία ευχαριστούμε. Όλα αυτά επέτρεψαν να προωθήσουμε τη συζητήσεις ε, σχετικά με τις προπτικές της συνεργασίας μεταξύ όλων των ε, Ευρωπαίων ε, εμπλεκομένων μετά από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Υπάρχουν και διάφορα παραδείγματα τα οποία αναφέρθηκαν και που αναφέρονται στο πρόγραμμα παραδείγματος χάρη της Πόλεως Λούμπλιν για τις χώρες της Ανατολικής Συμμαχίας όπου συζητήσαμε ε, την κοινωνία των πολιτών και τη συνεργασία με τη Λευκορωσία τονίζοντας πόσο σημαντική είναι η αλληλεπίδραση των πολιτιστικών προγραμμάτων στην κοινωνία των πολιτών και τον ρόλο του πολιτισμού ή στη διαδικασία εκδημοκρατισμού. Η, πολιτική η πολωνική προεδρία θα ήθελε να προωθήσει και την πολιτιστική συνεργασία και να την τονίσει. Γι' αυτό και έχουμε αναφέρει τη δυνατότητα η οποία υπάρχει στα πλαίσια μας να προωθήσουμε την πολιτιστική συνεργασία και αυτό ήταν ένα από τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν μαζί με ε, την ανατολική συνιστόσα της κινητικότητος που συζητήθηκε στο συνέδριο στη Βαρσοβία τον Ιούλιο. Ήρθαν πολλές, πολλές, ε, πολλοί εκπρόσωποι από τις γειτονικές χώρες και υπήρξε η δυνατότητα να προωθήσουμε ευρωπαϊκά προγράμματα για να προωθήσουμε την κινητικότητα. Αυτή λοιπόν η σύσταση τονίστηκε και πάλι το Σεπτέμβριο στο Συμβούλιο Υπουργών στην Βαρσοβία και η Δανική Προεδρία θα συνεχίσει αυτό το πρόγραμμα για να υπάρχουν συναντήσεις των υπευθύνων για τον πολιτισμό και των εκπροσώπων των Υπουργείων Εξωτερικών για να συνδυάσει κανείς πολιτισμό και διεθνείς σχέσεις. Αν σκεφτούμε λοιπόν πόσο κοντά είναι η μία, ο ένας πολιτισμός στον άλλων και πόσο ίσως αποκλίνουν οι προσπάθειές μας, τότε ε, θα γνωρίζουμε καλύτερα πώς να αντιμετωπίσουμε ε, τα τεκτενόμενα, όπως παραδείγματος χάρη εις ε, την Μεσόγειο, όπου η συνεργασία καθίσταται όλο και πιο σημαντική και πρέπει να πούμε εδώ ότι όλα αυτά θα πρέπει να συνδυαστούν με συγκεκριμένα μέτρα κατά τρόπον ώστε να έχουμε ε, εκτενή πολυσχηδή προγράμματα και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις οι οποίες υπάρχουν μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την σημερινή συνάντηση διότι πιστεύω ότι έτσι μπορούμε να προωθήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και πρέπει να σας πω ότι και εγώ διαπίστωσα λέει πρόεδρος στην Πολωνία πόσο η πολωνική η Προεδρία προσπαθεί να προωθήσει τα πολιτιστικά θέματα και επειδή έχουν τόσους γείτονες πιστεύω ότι θα μπορέσουν να επεκτείνουν τη δράση τους προς τις γειτονικές τους χώρες και στο τέλος του χρόνου δεν θα είσαστε πια στην Προεδρία του Συμβουλίου αλλά μπορείτε να προωθήσετε τη δράση σας στο τρίγωνο και ε, πιστεύω ότι και οι Δανείοι θα σας βοηθήσουν. Και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Σουσά, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όταν βλέπω εδώ τον κύριο Ντουζαρντάν, Θυμάμαι μία συνάντηση στην οποία είχα συμμετάσχει πριν από τρία χρόνια και ήταν συντονιστής της συζάτησης αυτής. Υπήρχαν πολύ σημαντικές προσωπικότητες στα πλαίσια του πολιτισμού στην Ευρώπη και ήταν παρόν και ο κύριος Μπαρόσο στη συνάντηση αυτή, ο πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και υπήρχε ένα ομόφωνο μήνυμα που ερχόταν από όλε αυτές τις προσωπικότητες προς τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το μήνυμα αυτό ήταν ότι η Ευρώπη διανύει μια κρίση, κύριε Πρόεδρε. Αυτό όμω το οποίο δεν διανύει κρίση, αυτό το οποίο παραμένει ιδιαίτερα ισχυρό, αυτό που είναι ένα από τα πιο πολιτικά, πολύτιμα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, τόσο στο εσωτερικό της Ευρώπης όσο και στο εξωτερικό της Ευρώπης. Έτσι λοιπόν η δυνατότητα της χρησιμοποίησης του πολιτισμικού δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι το οποίο θα απασχολήσει την Επιτροπή σας αύριο, κυρία Πρόεδρε, όταν ο Πρόεδρος μας θα έρθει να παρουσιάσει τη δική σας Επιτροπή το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συγχωρείτε, για την πρόθεση του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Και συζητάμε επίσης σήμερα τις δυνατότητες που έχει ο ευρωπαϊκός πολιτισμός να χρησιμοποιηθεί περισσότερο στα πλαίσια της εξωτερικής δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν αρχίσει να ελοποιούνται. Δεν θα αναφέρω αυτά τα οποία είπε εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης αναφέρθηκε σε ένα καταπληκτικό κατάλογο δραστηριοτήτων. Εγώ θα αναφερθώ σε κάποια πράγματα τα οποία ενδεχομένω δεν ακούσαμε ακόμα τις δραστηριότητες διεύρυνσης, τα πλαίσια της διεύρυνσης, με την υποστήριξη της ελληνική Διεύθυνσης Διεύρυνσης, την διαδικασία της Λουμπλιάνα, τη συνεργασία με τις υποψήφιε χώρες στα Βαλκάνια. Όλα αυτά είναι καταπληκτικά, φανταστικά. Η Καρολίνα αναφέρθηκε πριν από λίγα λεπτά στο πώς οι Προεδρίες Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχουν. Αναφέρθηκε στην Ουγγρική, την Πολωνική Προεδρία. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω ότι υπάρχουν κάποιες παρελθούσεις προεδρίες, όπως η Γαλλική Προεδρία του 2008, που κατέληξε συγκεκριμένα συμπεράσματα του Συμβουλίου για το ζήτημα αυτό. Να βερθώ επίσης στην ερχόμενη Προεδρία, την Δανική, η οποία θέτει την εξωτερική δράση στα πλαίσια, στην καρδιά της πολιτισμικής ατζέντα της Ένωσης. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά πράγματα τα οποία ήδη γίνονται. Για ποιο λόγο λοιπόν Μα ζητά ο κύριος Βάγνερ μια πρωτοβουλία για περισσότερη Ευρώπη. Για ποιο λόγο υπάρχουν, ε, έχουμε την κυρία Σάκη με την εξαιρετική αυτή έκθεση της Επιτροπής σας. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν μολονότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα ακόμα σε εξέλιξη, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να ακούσουμε περισσότερο την κοινωνία των πολιτών, που πάντα βρίσκεται κάποια βήματα μπροστά από μας. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να εξετάσουμε περισσότερο την καταπληκτική αυτή πρωτοβουλία, More Europe, και θα ήθελα να συγχαρώ τον Gottfried Wagner, καθώς επίσης και τα Ινστιτούτα που βρίσκονται πίσω από την πρωτοβουλία αυτή. Η πρωτοβουλία αυτή επιφέρει κάτι το πολύ σημαντικό στην όλη διαδικασία και συνοψίζοντα τα όσα ακούσαμε από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από του εμπειρογνώμονε, αν υπάρχει ένα σημείο στο οποίο όλοι συμφωνείτε, αυτό είναι το ακόλουθο κατά την άποψή μου. Χρειαζόμαστε μία στρατηγική, χρειαζόμαστε συνεργασία, χρειαζόμαστε συντονισμό, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ορατότητα, μεγαλύτερη προβολή. Νομίζω λοιπόν ότι στον τομέα αυτό θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε περισσότερο. Εδώ πρέπει να καλύψουμε τα κενά. Όλα τα στοιχεία αυτά είναι πολύ σημαντικά για το μέλλον και δεν αναφέρομαι μόνο στην επόμενη δεκαετία. Θα ήθελα να δω περισσότερες εξελίξεις στον τομέα αυτό του χρόνου. Μετά από δύο χρόνια το πολύ υπάρχουν πολλές προκλήσεις μπροστά μας αλλά και πολλές ευκαιρίες και θεωρώ ότι ε, η ευθυγράμμιση των όσων κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις πρωτοβουλίε τη κοινωνία των πολιτών και με την καταπληκτική έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με τα καταπληκτικά πορίσματα αυτής της ακρόασης, νομίζω ότι αυτό θα είναι σημαντική προτεραιότητα για μας. Αν καταφέρουμε να κάνουμε αυτό το θετικό άλμα, τα κρατη μελη του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς επίσης και οι οργανώσεις στα πλαίσια του πολιτιστικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Αν καταφέρουμε λοιπόν να συνεργαστούμε θα συμβάλλουμε πολύ στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης θα συμβάλλουμε πολύ και σε εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες. Αναφερόμενο σε αυτή την συνεργασία που έχουμε στο εξωτερικό, ναι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο soft power, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την, τον όρο πολιτιστική διπλωματία. Πέρα από αυτά, αυτό που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι οι αμοιβαίε ισότιμες ανταλλαγές. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μπορούμε και εμείς να μάθουμε από τις χώρες αυτές. Σαφώς μπορούμε να εξάγουμε κι εμείς, σαφώς μπορούμε να τους διδάξουμε πράγματα, αλλά έχουμε να μάθουμε ακόμα περισσότερα πράγματα από αυτούς, από τις, τρίτε από τις χώρες. Μόνον υπάρχει αυτή η αμοιβαία ισότιμη ανταλλαγή, τότε μόνο θα μας αντιμετωπίσουν σαν ισότιμο εταίρο, σαν αξιόπιστο εταίρο και μόνο τότε θα καταφέρουμε να κερδίσουμε και τον σεβασμό τους. Θα μπορούσαμε λοιπόν να επικεντρωθούμε στα σημεία αυτά και να συνεργαστούμε Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κράτη-μέλη καθώς επίσης και οι εκπρόσωποι του δημιουργικού τομέα και του πολιτιστικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ωραία. Φτάσαμε λοιπόν στο συμπέρασμα και η Προεδρία πάντα εξάγει τα συμπεράσματα. Σας ευχαριστώ όλους για, την, για τις γνώσεις σας, για την πραγματογνωμοσύνη σας, για τον τρόπο που πλησιώσατε τις ιδέες μας και επίσης ευχαριστώ που δεν ξεχάσατε τους καλλιτέχνες. Ε, συνεργαστήκατε και σας ενέπνευσαν. Είναι πολύ σημαντική η κοινωνία των πολιτών, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ποτέ τους δημιουργούς, τους καλλιτέχνες. Για την Ευρώπη και την ψυχή της Ευρώπης χρειαζόμαστε ε, να τους τοποθετούμε στον πυρήνα της συζήτησης. Τώρα έχουμε ακόμα δύο πρωτοβουλίες. Ε, έχουμε πολύ κόσμο που εργάζεται όχι μόνο στον τομέα του πολιτισμού αλλά και σε άλλους τομείς για να γίνει πιο ορατή και να προχωρήσει η Ευρώπη για να ξέρουμε τι σημαίνει τι είναι να είναι κανείς καλλιεργημένος, ποιος είναι πραγματικός άνθρωπος και αυτό δεν είναι γνωστό παντού με τον ίδιο τρόπο. Ευχαριστώ λοιπόν όλους την Προεδρία, τους συναδέλφους, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήσασταν πολύ περισσότεροι συνάδελφοι εδώ από όσους περίμενα και χαίρομαι που το κάναμε. Και θα ήθελα να κλείσω το σημείο αυτό. Μείνετε μισή ωρίτσα για να ανταλλάξουμε ε, απόψει με τα ευρωπαϊκά φεστιβάλ. Για να δούμε ποιος ε, μπορεί και όποιος θέλει να έρθει σε μεγαλύτερη επαφή με αυτούς τους φορείς. Όποιος δεν μπορεί να μείνει παρακαλώ να φύγει χωρίς να κάνει θόρυβο γιατί βιαζόμαστε. Σας δίνω λοιπόν δύο λεπτά για να βγείτε από την αίθουσα και θα συνεχίσουμε. Our final agenda item today is an exchange of views with Λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι η ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους η Ένωση Ευρωπαϊκών Φεστιβάλ ΕΦΑ που ε, είναι ένα δίκτυο διεθνές που δημιουργήθηκε το 1952 από την Denise de και θα ε, ε, εορτάσει η 60 ετία του χρόνου. Ε, εξετάζουμε λοιπόν ποιος είναι ο ο ρόλος του πολιτισμού και η ΕΦΑ είναι ένα ζωντανό παράδειγμα συσφίξεως μεταξύ των χωρών. Και τώρα υπάρχει η κυρία Κατρίν Τεβεντέ η οποία θα μας μιλήσει για την εργασία αυτής της οργανώσεως και της δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι, σας βλέπω που κάθεστε και πίσω μου. Το θέμα είναι ποιος είναι ο ρόλος του πολιτισμού στην κοινωνία μας και ποιος είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το πλαίσιο. Η δική μου παρέμβαση ήταν πολύ συγκεκριμένη για το πώς λειτουργεί ο κλάδος. Θα μιλήσω για τα φεστιβάλ στην Ευρώπη και το βασικό ερώτημα είναι πώς τα φεστιβάλ αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πιο αποτελεσματικό τρόπο, να απευθυνθούν σε, περισσότερο, σε μεγαλύτερο κοινό, σε επιχειρήσεις, σε άλλους φορείς και να κάνουμε τα φεστιβάλ ε, κινητήριο δύναμη για την Ευρώπη. Εκατο... Χιλιάδες ε, πολίτες επισκέπτονται τα φεστιβάλ και επιτρέπουν την πολιτική έκφραση σε συγκεκριμένο χρόνο, σε συγκεκριμένο μέρος, για την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Από τον Ίσνη, ε, Νόκορο, στο Ρίλ, από τον Μπέργεν στην Αθήνα, από το Μαυροβούνιο στις Βρυξέλλες. Σε όλα αυτά τα μέρη βρίσκεται κανείς ε, το κοινό σας και πρέπει να σας πω πως μόνο το 5% της Ένωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχει στη δημόσια συζήτηση για τα ευρωπαϊκά θέματα. Οι, ευρωπαϊκ... εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν όλο και μειωμένη συμμετοχή από το 62% το 79% στο 43% το 2009 η Ευρώπη φαίνεται πως έχει αφήσει πίσω τους πολίτες. Και στην πρόταση για, την, για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών το 2013 δεν υπάρχει καμία αναφορά στην πολιτική διάσταση και στη δυνατότητα που έχει να ε, δημιουργήσει ε, ένα μεγάλο κροατήριο, ένα μεγάλο κοινό. Παράδοξο αυτό. Πάντα ήταν μια διεθνής ε, πρακτική των δημιουργών και των καλλιτεχνών να ε, δημιουργούν διασυνοριακή κινητικότητα ε, με τη συμμετοχή τους στα πολιτιστικά δρόμενα και βέβαια με τον προγραμματισμό των φεστιβάλ. Ε, η μετανάστευση από εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μπορεί να έχει και μία πολιτική διάσταση. Και παρόλα αυτά φαίνεται πως η, εξωτερική, η ομάδα εξωτερικής δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τη Βαρόνη Άστον δεν έχει ακόμα ε, τμήμα ε, για τον πολιτισμό. Δεν είναι παράδοξο λοιπόν που η Ευρώπη ακόμα δεν έχει κάτι τέτοιο. Στα φεστιβάλ έρχονται άτομα από παντού. Ο διαπολιτισμικός διάλογος δεν είναι απλό σλόγγαν, είναι μια πραγματικότητα ε, που ε, γιορτάζεται στις εκδηλώσεις που γίνονται στις πόλεις, στους δρόμους, στις αίθουσες συναυλιών. Παράλληλα, έχουμε μια απίστευτη έκρηξη εθνικισμού, λαϊκισμού, ε, τάσεων που εναντιώνονται στην μετανάστευση, που συνδέονται βέβαια με τα μέτρα λιτότητα στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει συνέστημα, δεν υπάρχει αλληλεγγύη. Πού είναι η Ευρώπη. Υπάρχουν πάρα πολλά τεκμήρια για το οικονομικό αντίκτυπο των φεστιβάλ και των πολιστικών ε, φορέων ε, μια και τα φεστιβάλ δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξη. Το ξέρουμε. Επίσης, νέες μελέτες δείχνουν πως η έμεση ε, επίπτωση στην υγεία, στα κοινωνικές δεξιότητες και στην ε, ευεξία, ψυχική ευεξία είναι ακόμα περισσότερα από την άμεση ε, επίδραση, όπως μας είπε πρόσφατα στις Βρυξέλλες ο Πιέρ Λουίτζι Σάκο. Η ατζέντα του 2020 για την ευφυή βιώσιμη ε, ανάπτυξη για όλους είναι μια στρατηγική στην οποία πρέπει να ψάξει κανείς πολύ να βρει τη διάσταση του πολιτισμού και δεν αναφέρεται ρητά. Ακολουθούμε αυτές τις τάσεις στην Ευρώπη. Τα φεστιβάλ φέρνουν τα μεγάλα ονόματα των δημιουργών στη σκηνή και επειδή τα ε, ΜΜΕ ασχολούνται με τα φεστιβάλ, τα μηνύματα μπορούν να αγγίξουν μεγάλο κοινό, νέο και ηλικιωμένο. Και στα διοικητικά του συμβούλια έχουν εκπροσώπηση των τοπικών επιχειρήσεων και των τοπικών ε, πολιτικών. Έτσι ε, συναντιόνται για δεξιώσεις, για εκδηλώσεις και κάθε μέρα έρχονται σε επαφή με τους διευθυντές των φεστιβάλ. Και παράλληλα στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες ψάχνουν με νέες μορφές εταιρικής σχέσης με τις επιχειρήσεις και ψάχνουμε ε, κάποιους τους καινούριους ηγέτες που θα μας εκφράσουν, ε, που λείπουν, ε, που πρέπει ε, από κάποια σκηνή να φέρουν τη φωνή τους στο κοινό. Γιατί λοιπόν να μην χρησιμοποιήσει η Ευρώπη τα φεστιβάλ. Τα φεστιβάλ καλωσορίζουν χιλιάδες καλλιτέχνες στη σκηνή και είναι καινοτόμα, δημιουργικά και αυτό μας το έδειξε και το Ευρωπαϊκό Έτος του 2009. The objectives defined in... Και οι στόχοι που έχουμε ε, στην ατζέντα μας δεν αναφέρεται στην ε, πολιτιστική δραστηριότητα. Για ποιο λόγο. Αφού το πρόγραμμα για τη Δημιουργική Ευρώπη, ε, εξ όσο γνωρίζουμε, συμπεριλαμβάνει και τη δημιουργική βιομηχανία, όπως επίσης και την πολιτιστικό μη κερδοσκοπικό κλάδο. Θα πότε θα επενδύσει λοιπόν στις δημιουργικές δεξιότητες αυτού του κλάδου η Ευρώπη. Γιατί ας μην ξεχνάμε πως υπάρχει ο πολιτισμός και η βιομηχανία του πολιτισμού. Θέλουμε λοιπόν ένα πραγματικό πρόγραμμα για τον πολιτισμό. Αυτή τη στιγμή 800 τουλάχιστον φεστιβάλ ζητάνε επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και πρέπει να δούμε στο ευρωπαϊκό πλαίσιο τι γίνεται. Υπάρχουν πολλά φεστιβάλ, αλλά όχι όλα είναι επιτυχημένα. Κάποια έχουν τόσο χαμηλό, ε, χαμηλές επιδόσεις που θα έλεγα πως μόνο το 8% έχει κάποια οικονομικά θετικά αποτελέσματα. Θέλουμε λοιπόν μια ανοιχτή κοινωνία, μια κοινωνία που ευημερεί, αλλά δυστυχώς η γνώση που έχουμε για τον πολιτισμό δεν φαίνεται στις κοινωνίες μας και βέβαια αυτό που κάνουν είναι μια πολύ απολυστευμένη παρουσίαση δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε παρανοήσεις. Ξέρουμε πως ο πολιτισμός δεν μπορεί να λύσει όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα δεν θα έπρεπε να ε, υποκαταστήσει ε, την πολιτική, αλλά το ακούσαμε σήμερα το απόγευμα. Θα πρέπει να κατανοήσουμε μαζί πόσο δυνατές είναι οι τέχνες και ο πολιτισμός της κοινωνίας μας και τι μπορεί να κάνει για τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ο πολιτισμός, όπως βέβαια και το τι δεν μπορεί να κάνει. Οπότε έχουμε τέσσερις ερωτήσεις, τέσσερις ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσουμε. Ποιος, ποιοι είναι οι πολιτική για τα φεστιβάλ στην Ευρώπη. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ε, συνθήκες για να ανθούν τα φεστιβάλ. Δεύτερον, πώς μπορούμε να ε, χρησιμοποιήσουμε το πλεονέκτημα που προσφέρουν τα φεστιβάλ. Τρίτον, πώς μπορεί η προσέγγιση αυτή των φεστιβάλ να γίνει μια δημιουργική δύναμη για την Ευρώπη. Εκατοντάδες παντού, σε όλες τις πόλεις, σε όλες τις περιφέρειες. Και τέσσερα, μια και είναι τόσο Ποιος είναι ο ρόλος πια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ. Για να ε, δούμε για ένα λεπτό ποια είναι τα βασικά σημεία κίνησης για κάθε ε, πολιτιστική δραστηριότητα και πολιτική. Ποιος είναι ο ρόλος του καλλιτέχνη στην δημιουργία. Κάθε πρόγραμμα θα πρέπει να δίνει όπλα ε, στον καλλιτέχνη για να αναπτυχθεί δημιουργικά και ελπίζω να μην να μην μας κορυδεύει η ιστορία, όπως μας είπε ένας πολύ πετυχημένος επιχειρηματίας από την Αυστραλία. Να μην πούμε εμείς, ε, να μην πούνε κάποτε πως ο αιώνας μας έκανε μια χρηστική προσέγγιση στην τέχνη, όπου το μόνο που μετράει είναι ο αριθμός του κοινού, οι στατιστικές στον τουρισμό και τα δικαιώματα copyright ε, για ε, όσα που θα πρέπει να αποτελούν ένα χώρο σκέψης, πειραματισμού και δημιουργίας. Ας εξασφαλίσουμε, είπε αυτοί οι επιχειρηματίες, πώς θα εξυπηρετήσουμε τους καλλιτέχνες και θα ε, ενδυναμώσουμε τα δικαιώματά μας. Έχουμε ευθύνες ε, προς το κοινό και προς τους καλλιτέχνες. Και τα φεστιβάλ θα πρέπει να κάνουν καλές επιλογές και να μας δώσουν τροφή για σκέψη, να μας εκπλήξουν, να σπρώξουν τα όρια μας. Στην ε, ε, στην πραγματικότητα είπε ο διευθυντή του Φεστιβάλ τη Αβενιών πως θα πρέπει το φεστιβάλ να ορίζει κάποιες εκδηλώσεις που προωθούν την καινοτομία, τη δημιουργικότητα. Ο ρόλος του φεστιβάλ είναι να επιτρέψει στους καλλιτέχνες να ξεκινήσουν κάποιες δραστηριότητες οι οποίες δεν θα μπορούσαν να κάνουν μέσα από κάποιους άλλους φορείς. Και το δεύτερο σημείο κίνησης είναι πως για κάθε πρόγραμμα θα πρέπει να ζητήσουμε από τα φεστιβάλ να ανταποκριθούν σε αυτές τις υποχρεώσεις. Και πριν φτάσω στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να σας δώσω ένα παράδειγμα από φεστιβάλ που είχαν κάποια πρωτοπόρα δράση στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Είναι ε, η, Ένωση για τα Ευρωπαϊκά Φεστιβάλ. Το 1952 ο Ίγκορ Μάρκεβιτς ε, και ο Ντεμίντε Ρουσμό ε, ίδρυσαν αυτή την ένωση. Είναι η παλαιότερη ένωση που εκπροσωπεί πάνω από 111 φεστιβάλ στην Ευρώπη. Και θέλουμε η διασυνοριακή συνεργασία από το ευρωπαϊκό στο τοπικό επίπεδο, από τα φεστιβάλ από την Ευρώπη να απαντήσει και το ποιο θα είναι ο ρόλο Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί βέβαια τα χρήματα πάντα θα είναι λίγα. Ε, Όμω δεν θα πρέπει να είμαστε υπερβολικά μετρημένοι στι προσπάθειέ μα. Έχει την αρμοδιότητα η Ευρώπη. Μπορεί να εξασφαλίσει την πολιτιστική πολυμορφία τη Ευρώπη και θα δώσει την αίσθηση του ανήκειν στου Ευρωπαίου πολίτε. Δεν θα πρέπει να αφήσουμε στην τύχη τη τον πολιτισμό. Δεν θα πρέπει να αφήσουμε τον εθνικισμό να μας κατακτήσει. Ε, η ερώτηση που πρέπει να απαντήσουμε είναι όχι πώς μόνο θα σώσουμε την Ευρώπη, αλλά το πώς θα αποκριθούμε στο γιατί και το διότι του ε, πώς σώζεται η Ευρώπη. Νομίζω πως τα φεστιβάλ μπορούν να γίνουν πιο αποδοτικά, να ε, τα χρησιμοποιήσουμε στη διαδικασία εκδημοκρατισμού μεγαλύτερου οικοδομικοσμού τη Ευρώπη. Και έχω ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, τα φεστιβάλ για την Ευρώπη, η Ευρώπη για τα φεστιβάλ. Ένα πρόγραμμα που θέλει να έχουμε περισσότερα φεστιβάλ Γιατί... Its aim is to... προώθηση της Ευρώπης και του πολιτισμού. Για να έχουμε μια θετική ενέργεια με τα εκατοντάδες φεστιβάλ που πάρα πολλά ζητούν επιχορηγήσεις και πολύ λίγα λαμβάνουν. Ένα νέο πρόγραμμα που θα δίνει στα φεστιβάλ ε, τη δυνατότητα να αποτελέσουν τμήμα της διαδικασίας ολοκλήρωσης της υπήρους μας. Και εδώ έχουμε διάφορα στοιχεία. Ε, το βασικό είναι να έχουμε ένα εγχειρίδιο ε, το οποίο θα ε, είναι σε βιβλίο, θα είναι εφαρμογή και θα είναι και ιστότοπος. Και κάθε δεύτερο χρόνο έχει δύο ομάδες στόχο που είναι το, η σήμανση που λέει Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ και βέβαια ένα βραβείο του Φεστιβάλ για την Ευρώπη που δίδεται μόνο σε κάποιο μικρό ρυθμό φεστιβάλ. Θα δώσει πολλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα Βελιγάστα. Θα ξεκινήσει με λίγα και πολλά από αυτά τα φεστιβάλ θα γίνουν τμήμα της δυναμικής διαδικασίας. Τοπικά δίκτυα, τοπικοί συνεργάτες που θα δίνουν αυτή την ε, σήμανση και θα συμπεριλαμβάνει και τα εμβληματικά φεστιβάλ, όπως επίσης και τα πολύ μικρά που ασχολούνται με συγκεκριμένα πολύ κλειστά θέματα. Θα δώσει μια μεγαλύτερη ορατότητα στα φεστιβάλ και επιπλέον αυτά τα φεστιβάλ θα γίνουν πιο γνωστά στην Ευρώπη και η Ευρώπη θα, κάνει, θα γίνει πιο γνωστή στους πολίτες μέσω των φεστιβάλ. Λοιπόν, θα πρέπει να πω, επειδή γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή συζητιέται προπολογισμό στην ε, ε, Ευρω... στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Ξέρουμε τι θα παρουσιαστεί αύριο εδώ. Θα σας ζητήσω, κύριοι Ευρωβουλευτές, να κάνουμε μια κοινή έκκληση για ένα ε, πειραματικό σχέδιο για τα φεστιβάλ που θα προωθεί στα φεστιβάλ μαζί με την Ένωση για τα Ευρωπαϊκά Φεστιβάλ. Και υπογραμμίζουμε την πρόθεσή μας να στηρίξουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον πολιτισμό, στον προϋπολογισμό που προτείνει και θέλουμε εδώ ε, να έχει μια μεγάλη να έχουμε μια μεγάλη στήριξη κυρίως στο, στις μη κερδοσκοπικές ενώσεις και δημιουργούς. Θέλουμε επίσης μια μεγαλύτερη αναγνώριση των τεχνών και των δημιουργών στα διαφορετικά ταμεία και στα περιφερειακά ταμεία. Και τέλος, προτείνουμε στα, στους ε, βουλευτές να πάνε στα φεστιβάλ και να έρθουν σε συζήτηση με τους ε, ε, τοπικούς δημιουργούς και με τα Υπουργεία σε τοπικό επίπεδο για να στηρίξουν τον πολιτισμό. Γιατί βέβαια εδώ είμαστε αρμόδιοι για πολλά πράγματα, αλλά την αρμοδιότητα για τα φεστιβάλ τα έχουν οι τοπικοί παίκτες και σας καλούμε βεβαίως και κλείνω στην 60, στον 60ο εορτασμό της Ένωσης που θα εορτάσουμε στον Μπέρκεν της Νορβηγίας Νορβηγίας με τίτλο ε, «Εόρτασε τις, ε, «Γιόρτασε τις τέχνες, γνώρισε τον κόσμο ε, και χαίρομαι που μένουν και λίγα λεπτά για να μου υποβάλλετε ερωτήσεις. Θα σας μοιράσω βεβαίως και κάποια γραπτά κείμενα μετά την λήξη συνεδρίασης για να είστε περισσότερο ενήμεροι. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Βέβαια, περάσατε πολύ γρήγορα και ελπίζω όλοι να σας κατάλαβαν. Ε, θα υπάρξει ένα πρόγραμμα για την Ευρώπη το οποίο έχω ήδη υπογράψει. Σας υπενθυμίζω διότι είναι εδώ όλοι οι συντονιστές ότι του χρόνου για το νέο δημοσιονομικό έτος χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα πιλωτικό ε, η Ευρώπη για τα φεστιβάλ και τα φεστιβάλ για την Ευρώπη και θα συναντήσουμε εκεί ανθρώπους που δεν συναντούμε πουθενά αλλού και τους οποίους θα μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε για το πρόγραμμά μας, για το όραμα του Ρομπέρ Σουμάν. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική ιδέα την οποία έχουν εκπονήσει ε, οι συνεργάτες και θα πρέπει να την προωθήσουμε. Σήμερα δεν θα προλάβουμε. Δεν νομίζω ότι κανείς συνάδελφος θα τολμήσει κάτι να ρωτήσει γιατί τελειώσαμε. Αλλά ευχαριστώ την Κατρίν και τους συνεργάτες και θα το δούμε πολύ σοβαρά και τουλάχιστον στον επόμενο προϋπολογισμό και στην συζήτηση του πολιτιστικού προγράμματος θα ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση για να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε. Σας ευχαριστώ και σας και τους υπολείπους και έτσι ολοκληρώθηκε η ημερήσια διάταξη και πάμε στην συνεδρίαση των συντονιστών. Οι υπόλοιποι μπορούν να φύγουν και να περάσουν καλό βράδυ.